Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή αυτή συνεδρίαση της μαραθώνιας συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών. Συνεδριάσαμε και χθε και σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμανς, για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας στα πλαίσια του διαρθρωτικού διαλόγου. Έχουμε λοιπόν τον δικό μας επίτροπο που αφοσιώνεται στο έργο της Επιτροπής Αναφορών με κοινέ αξίες όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους ανησυχίες και προβλήματα προσπαθώντας να τα επιλύσουμε. Πολλά κοινά λοιπόν έχουμε μεταξύ μας. Θέλω επίσης να σας πω ότι η τάση στην Επιτροπή Αναφορών αυτή την εποχή είναι το περιβάλλον. Είναι επίσης τα δικαιώματα των παιδιών, ε, το δικαίωμα ε, στις εκλογές, το εκλέγιν. στις εθνικές εκλογές των ε, χωρών τους και των χωρών κατοικίας τους. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία. Τώρα βλέπετε με το δημοψήφισμα προέκυψαν διάφορες σχετικές αναφορές. Οι εκλογικοί νόμοι επίσης απασχολούν την ε, Επιτροπή μας τελευταία. Έχουμε και αναφορές κάποιες τουλάχιστον για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα νέο θέμα για την Επιτροπή μας από το 2015. Και σχετίζονται βέβαια με τους πολυάριθμους ε, μετανάστες που έχουν φτάσει στις ακτές μας. Σε σχέση λοιπόν τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσείς έχετε πει ότι θα παίρνω απάντηση ενδιαφέροντα σε τρεις μήνες και είναι κάτι που δεν έχουμε πετύχει ακόμα απόλυτα, αλλά προσπαθούμε. Θέλω να τονίσω ότι είσαστε φρόσδεκτος στην Επιτροπή μας για να μας σχολιάσετε ό,τι έχετε να μας πείτε από πλευρά Επιτροπής. Παρακαλώ. Τίμερμανς, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και τότε στην τελευταία χρονιά τόσα πολλά έχουν επιτευχθεί και ευχαριστώ πολύ τη δικιά σας Επιτροπή και σας όλους ιδιαίτερος κυρία Πρόεδρε που πραγματικά ενισχύσατε το έργο της Επιτροπής αυτής και συνεργαστήκατε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπατε και εσείς δεν έχουμε συμμορφωθεί ακόμα πλήρως με τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει να απαντάμε σε κάθε αναφορά μέσα σε τρεις μήνες, αλλά κοντεύουμε. Και θα γίνει. Ελπίζω πάντα. Μερικέ φορέ καταλαβαίνετε ότι οι αναφορέ αναφέρονται σε ζητήματα που είναι αρκετά δύσκολα και περίπλοκα. Τώρα γιατί η Επιτροπή Αναφορών και το έργο της είναι τόσο σημαντικά για μένα. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι ένα από τα λίγα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να έχουμε απευθείας επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες για θέματα για τα οποία έχουν άποψη, για θέματα που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τα δικαιώματά τους και παρόλο που βέβαια πρόκειται για ατομικέ αναφορές, αν τις εξετάσετε γενικότερα, ίσως θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο μοντέλο που ακολουθούν και που ίσως να μην έχουμε, να μην μπορούσαμε να είχαμε καταλάβει αν δεν είχαμε τις αναφορές. Εγώ έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις που το αποδεικνύουν αυτό. Ότι υπάρχουν κάποια επαναλαμβανόμενα θέματα. Όπως είπατε για το περιβάλλον. Είναι ένα παράδειγμα. Η περίφημη ιστορία του αεροδρομίου στη Γαλλία. Μπορούμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη Γαλλία να αποφύγει λάθη, σφάλματα. Και αυτό γίνεται ακριβώς επειδή Μα στάνουν αναφορές για τέτοια θέματα. Τώρα υπάρχουν άλλοι τομεί που για μένα προσωπικά έχουν μεγάλη σημασία και που έχουν να κάνουν με το έργο σα. τα δικαιώματα, ε, θεμελιώδη δικαιώματα, η διαφάνεια, περιβάλλον. Αν μπορώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας ε, ζητήσω να ενημερώνετε όλους εκείνους με τους οποίους είσαστε σε επαφή, να ξέρουν ότι υπάρχει το μητρό μας με διαφάνεια και ελπίζω να πετύχουμε συμφωνία τα τρία θεσμικά όργανα, ώστε να έχουμε όλο και περισσότερη διαφάνεια στο έργο μας. Αν μπορείτε, διαδώστε το αυτό. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας. Πράγματι είμαι ο δικός σας επίτροπος. Να είμαστε σε επαφή. Αν βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημερώστε με. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Βέβαια, πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε αναφορές για τις οποίες δεν διαθέτουμε νομικά μέσα για να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για να τις αντιμετωπίσουμε. Κάτι το οποίο βέβαια απογοητεύει πολύ τους αναφέρονται συχνά. Γιατί αν έχετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα δεν θέλετε να έρθει κάποιος από τις Βρυξέλλες και να σας πει «Α, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, είναι οι χώρες μέλη». Χάσατε. Συχνά όμως συμβαίνει, αλλά ακόμα και τότε μπορούμε κι εσείς κι εμείς να έρθουμε σε επαφή με τις χώρες μέλη και να προσπαθήσουμε να λύσουμε τέτοια ζητήματα, όπως ο εκλογικό νόμος είναι εθνική αρμοδιότητα βέβαια. Δεν είναι ευρωπαϊκή. Αν όμως διαπιστώνουμε ότι επίμονα παίρνουμε αναφορές για τη χρήση των γλωσσών ή για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχουμε διάλογο με την χώρα μέλος για να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Αυτά. Περιμένω τις ερωτήσεις σας τώρα και τα σχόλιά σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι συντονιστές πρώτα και μετά οι υπόλοιποι ευρωβουλευτέ, εφόσον έχουμε χρόνο μέχρι τις 4. Να είσαστε σύντομοι παρακαλώ. Πίτερ, εσείς πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ήσασταν σαφέστατος, είστε ο δικός μας Επίτροπος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Από την πρώτη και όλα στιγμή είστε κοντά μας και θέλω να πω ότι από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας η συνεργασία μας έχει γίνει πολύ καλύτερη και χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά όταν έχουμε έναν τόσο συνεργάσιμο συνομιλητή που μπορούμε να, ε, του, να μοιραστούμε μαζί του τις ανησυχίες μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Η επικοινωνία ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη ε, έχει βελτιωθεί, έχουν τηρηθεί αρκετά χρονοδιαγράμματα. Ε, εγώ προσωπικά έχω το εξή πρόβλημα. Όταν λαμβάνουμε απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλές φορές ε, χαρακτηρίζονται από ασάφεια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει η Επιτροπή. Γι' αυτό θα μπορούσαν ίσως ε, να σημειωθούν βελτιώσεις εδώ και θα μπορούσαμε ε, ίσως να σας ε, μεταδίδουμε καλύτερα τα ερωτήματα τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι έτσι θα αποφύγουμε καθυστερήσεις και υπερβολική γραφειοκρατία. Όταν κάτι έρχεται από την Επιτροπή, εμείς το θεωρούμε ασαφές και το ξαναστέλνουμε πίσω σε εσά. Μετά, θα επιθυμούσα να υπάρχει κοινή συμφωνία για τις ε, παραδεκτές και μη παραδεκτές αναφορές, δηλαδή συμφωνία μεταξύ ε, ημών τη Επιτροπής και ημών τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Γραμματείας, διότι πολύ συχνά έχουμε πρόβλημα με αναφορές οι οποίε ε, για μα είναι παραδεκτές, για εσά όχι και ούτω καθεξής. Σίγουρα οι αναφορές αντιμετωπίζονται με τον ίδιο δίκαιο τρόπο, όμως υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις τις οποίες διαφωνούμε κάθετα. Επίσης, θα ήθελα να συζητήσουμε το θέμα της διαδικασίας υπαραβάση και να ενημερωνόμαστε καλύτερα γι' αυτό, διότι έχουν παρατηρηθεί κάποια μικρά προβλήματα στην επικοινωνία εκεί. Έπειτα, κύριε Επίτροπε, πολλές φορές διατυπώνονται από την Επιτροπή μας επιθυμίες για αλλαγή, τροποποίηση της νομοθεσίας. Και εδώ θα επιθυμούσα μια ε, καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Θα μπορούσε, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, γίνεται περισσότερο ακουστό στις επιθυμίες αυτές από την Κομισιόν. Υπάρχουν, ε, υπάρχει ανάγκη για έναν καλύτερο και δίκαιο διάλογο. Σας ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, που ε, μίλησα περισσότερο από όσο μου είχατε επιτρέψει, αλλά υπήρχαν βασικά ερωτημάτα τα οποία έπρεπε να ε, θέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βεσερίλη από τους ε, S&T. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς που είσαστε εδώ και πάλι μαζί μας. Θα σας ρωτήσω μερικά συγκεκριμένα πράγματα. Δύο από αυτά έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία ακούσαμε ήδη. Δηλαδή πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, να ανταποκριθούμε στις καταγγελίες τους, γιατί μερικές φορές πλήττονται εξαιτία της περιοριστικής ερμηνείας του άρθρου 51 ε, της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολλέ οι αναφορές που μας έρχονται όσον αφορά την παραβίαση δικαιωμάτων, όπως είπαμε. Κάποιες έχουν να κάνουν με τη χρήση των γλωσσών ε, στις διάφορε χώρες, μάλες με τον ε, εκλογικό νόμο, όπως στη Βουλγαρία, που μόνο στη βουλγαρική γλώσσα υπάρχουν ε, κατάλληλοι κτλ. Και άλλες φορές περιορίζεται η ελεύθερη έκφραση ή το δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν πληροφορίες σε μια γλώσσα που κατανοούν και κυρίω όταν πρόκειται να συμμετάσχουν σε εκλογέ και να αποφασίσουν ποιο θα του κυβερνήσει. Έπειτα, 30 εκατομμύρια Ευρωπαίοι περιμένουν να υπογραφεί σε θήκη Μάρακετ για τα άτομα με μειωμένη όραση. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εμποδίζουν την κύρωση. Τι στρατηγική θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Και στο γενικότερο πλαίσιο της ερμηνείας του άρθρου 51 πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει ευρύτερη ερμηνεία έτσι ώστε να μπορούμε σωστά από πλευρά της Επιτροπής μας να δώσουμε την δέουσα προσοχή στις αναφορές των πολιτών. Και κάτι ακόμα για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Υπάρχει ένα υπερεθνικό φαινόμενο που είναι η τρομοκρατία των τζιχαντιστών. Εσείς ο ίδιος την ε, προηγούμενη εβδομάδα στις 14 Απριλίου όταν εγκρίναμε την οδηγία PNR είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, ότι πρέπει αποτελεσματικά να ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε, οι αρχές πληροφοριών δηλαδή για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Είναι ένα πρώτο βήμα για ανταλλαγή Όντω ε, στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών μελών και συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος που έλεγε ότι όλα τα μέτρα πρέπει να οδηγήσουν σε ένα σύστημα ε, κοινή υπηρεσία πληροφοριών μέσω μηχανισμών μεταξύ άλλων του δικτύου για την καταπολέμηση της σπαστικοποίησης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σολεδά καμπεθών. Ευχαριστώ. Δεν ήμουν εδώ από την αρχή, λυπάμαι. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που είναι μαζί μας και μπορούμε έτσι να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχω την αίσθηση ότι πάντα τον ε, υποδεχόμαστε καλά, μας ενημερώνει. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Λοιπόν, οι ερωτήσεις μου τώρα. Έχουν να κάνουν με το έργο της Επιτροπής Αναφορών, προφανώς. Κάποια πράγματα τα έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επιμένω γιατί επανέρχονται συνεχώς. Πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε μια διαδικασία ποιότητας και τι εννοώ, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η απάντησή μα στους αναφέροντε, γιατί πρέπει να συμμετέχουν εδώ όλα τα θεσμικά οργάνα, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρειαζόμαστε λοιπόν τη συμμετοχή και τη επιτροπή που συμμετέχει, αλλά και των χωρών μελών. Πρέπει δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε έγκαιρα απάντηση στους αναφέροντε με σωστέ πληροφορίε. Τι διαδικασία θα μπορούσαμε να έχουμε για να υπάρχουν εγγυήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι για την καλύτερη ρύθμιση που συζητάμε αυτή την εποχή, καλύτερη νομοθετική ρύθμιση, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς το βάζουμε, θα μπορούσε να το βάλει και η Επιτροπή. Από την αρχή της θητείας αυτής τώρα το συζητάμε το θέμα των αρμοδιοτήτων που έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που οι πολίτε πρέπει να το γνωρίζουν και εμεί να γνωρίζουμε έτσι ποιε αναφορέ είναι παραδεκτέ και ποιε όχι. Μερικέ φορέ υπάρχει ελαστικότητα. Θέλουμε έτσι καλώ να ακούμε όλου του πολίτε, όμω πρέπει να δίνουμε και απάντηση. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ευρύ πεδίο, να τους ακούμε όλους, αλλά να είναι και ξεκάθαρο πού έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού όχι. Τέλος, για το θέμα των παιδιών. Εδώ και ένα χρόνο δουλεύουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είδαμε ότι πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς προστατεύονται τα παιδιά, πώς προστατεύονται τα δικαιώματά τους τα παιδιά νομικά δεν έχουν τη δυνατότητα, ίσως δεν έχουν καν τα μέσα να προσφύγουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα ίδια. Αλλά είναι ένα τομέα αυτός που πρέπει να εξετάσουμε και ρωτάω, υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορούν να μπορούμε να δώσουμε φωνή στα παιδιά, όχι μόνο εδώ στην Επιτροπή Αναφορών, δεν εννοώ απαραίτητα αυτό, αλλά κάποιο τρόπο να βρούμε ώστε να δώσουμε φωνή στα παιδιά. Ευχαριστούμε κυρία Όκεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κύριε Τίμερμανς. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ε, βρίσκω εδώ και σας έστειλα και εγώ κάποιες, ε, μια επιστολή σχετικά με ένα θέμα, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες εδώ. Ε, πάντως, από ό,τι μαθαίνω στις κάτω χώρες, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με τη χρήση των μικρών πλαστικών σακούλων. Ωστόσο, το θέμα που είναι πολύ βασικό για μένα είναι η καλή διοίκηση, η χρηστή διοίκηση και ιδιαίτερα στα πλαίσια του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Εδώ παρατηρείται μια σύγκρουση συμφερόντων και πιστεύω πως απέχουμε πολύ ακόμα από το να καταφέρουμε να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα χωρίς συγκρούσει συμφερόντων. Βλέπω ότι υπάρχει μια αυξητική ε, τάση για αυτό το θέμα στην αίμα και αν πηγαίνατε κι εσείς εκεί θα βλέπατε ότι υπάρχουν ολοένα και ισχυρότεροι σύνδεσμοι ανάμεσα στην Έμα και στην βιομηχανία. Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι δεν αρκεί μία δήλωση ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εσείς και εγώ πρέπει να βρούμε λύσεις. Για να μην υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων και πιστεύω πως πρέπει οι απόψεις μας ε, να ε, συγκλίνουν και πρέπει να δείξουμε πυγμή και αποφασιστικότητα. Να μην δεχτούμε καμία απολύτως σύγκρουση συμφερόντων, ε, ιδιαίτερα στην διοίκηση και να καταστεί αυτό σαφέ. Μας αναφέρατε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασίας που αφορά την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. σχετικά με την, ε, που σχετίζεται και με τη σύμβαση περί διαφάνειας. Ωστόσο, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με την αποθεσία. Κινείται η κατάσταση. Οι πολίτες ε, θα μπορούν να δουν ότι τους παίρνουμε στα σοβαρά. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αλμπιόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω για ζητήματα που έχουμε εξετάσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Το ένα είναι η Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών, το TIP-TIP, όπου εμείς καταδικαίλουμε ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Πιστεύω ότι είναι πολύ ανησυχητικό και εδώ στην Επιτροπή αυτή που δίνουμε φωνή στους πολίτες, τουλάχιστον έτσι πρέπει να κάνουμε, όταν κάποιοι πολίτες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκουν μπροστά τους ένα τείχο. Πάνω από 3 εκατομμύρια υπογραφές μαζεύτηκαν σε πρωτοβουλία πολιτών και οι πολίτες αρνούνται τη συμφωνία αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω, ο κύριος Τίμερμανς γνωρίζει κατά πόσο θα αλλάξει κάτι ώστε να μπορούμε πάντα να τα αποκρινόμαστε στους πολίτες όταν αυτοί διαμαρτύρονται για κάτι. Δεύτερον, πολλές αναφορές έχουμε για πολίτες οι οποίοι απελούνται, για παράδειγμα, απελάθηκαν πάνω από 4.000 κοινοτικοί υπήκοοι μεταξύ αυτών πολλοί Ισπανοί από το Βέλγιο. Εδώ παραβιάζεται η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Γιατί ένα από τα λίγα καλά που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η ελεύθερη διακίνηση. Διακίνηση και η επιλογή κατοικίας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και τέλος, για το θέμα των αρμοδιοτήτων. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί η απάντηση που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα και άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όμως η ερώτηση είναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα όταν συστήνει στις χώρες μέλη να κάνουν περικοπές σε κοινωνικές πολιτικές, στην υγεία, την εκπαίδευση, στις συντάξεις. Όταν όμως οι περικοπές αυτές που συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τότε λέτε ότι δεν έχετε αρμοδιότητα. Για παράδειγμα, χθε συζητήσαμε εδώ για την πρόσβαση στην κατοικία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών η πολιτική κατοικία. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία υποχρέωσε την Ελλάδα, για παράδειγμα, να αλλάξει τον νόμο της, ώστε να μπορούν να γίνονται εξώσεις από την πρώτη κατοικία των ανθρώπων. Λοιπόν, τι γίνεται με τι αρμοδιότητε. Άλλοτε έχετε, άλλοτε δεν έχετε. Για περικοπέ έχετε, αλλά για να υποστηρίξετε τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Ακούσαμε πέντε ομάδε. Εσεί τώρα. Για να απαντήσετε, κύριε Τίμερμαντ. Δεν θα απαντήσω Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, θα προσπαθήσω σύντομα. Αν δεν είναι πλήρε οι απαντήσεις μου, τότε προτείνω να μας το πείτε. Να πείτε στην Επιτροπή δεν είναι πλήρη η απάντησή σας. Κάθε φορά δηλαδή που δεν δίνουμε πλήρε απαντήσει να μας το λέτε. Και αν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση θα το κάνουμε. Μπορούμε να έχουμε διάλογο με την γραμματεία σας για να το βελτιώσουμε. Αλλά θα το κοιτάξω. Αν δεν είναι πλήρε απαντήσει μα, εγώ θα το κοιτάξω. Γιατί βλέπετε είμαστε τόσο κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο του να απαντάμε έγκαιρα, που εννοείται ότι θέλουμε και οι ερωτήσεις να απαντούνται πλήρως. Οπότε θα δω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Για το τι είναι παραδεκτό και τι όχι. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα είναι ξεκάθαρο το ζήτημα αυτό. Η δικιά μου στάση είναι ότι αν ιδίω αν πρόκειται για ατομική περίπτωση, αν κάποιο φτάνει στο να σας στείλει αναφορά. Εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς και θα ήθελα να είμαι εντελώς ξεκάθαρος και να είναι σαφές για μένα κατά πόσο είναι κάτι παραδεκτό ή όχι. Ιδίω όταν πρόκειται για ατομικές περιπτώσεις. Γιατί με κάθε σεβασμό στην κυρία Ομπιόλ, κάποια από αυτά τα ζητήματα τα οποία υποβάλλονται ως αναφορές έχουν από πίσω τεράστιες εκστρατείες με χιλιάδες χιλιάδες ίδιο ακριβώς κείμενο που μας ήταν αναφορές δηλαδή με αντιγραφή του ίδιου κειμένου. Ε, τι σημαίνει αυτό. Αν οργανώνεται τόσο γρήγορα κάτι, ε, τότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα περισσότερο πρέπει να είμαι πιστός στους κανόνες από όταν είχα ατομικές περιπτώσεις όπου κανείς δεν έχει πουθενά αλλού να απευθυνθεί. Αν για το TTIP ή για άλλα έχετε χιλιάδες και χιλιάδες αναφορές, βεβαίως και τις παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι το πλαίσιο είναι διαφορετικό σε μια τέτοια περίπτωση από ότι στην περίπτωση κάποιου μεμονωμένου ατόμου ο οποίος ζει δίπλα σε ένα αεροδρόμιο και βλέπει εκεί να αλλάζουν τα πράγματα, οπότε αρχίζει και να ρωτιέται τι θα γίνει με την περιουσία μου, τι γίνεται με το περιβάλλον. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι για μένα τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Θα έλεγα ότι κάθε φορά υπάρχει ανθρώπινη διάσταση που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Αυτοί που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση σε μεγάλες εκστρατείες, σε μεγάλες οργανώσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους. Αυτή είναι η διαφορά μιας αναφοράς από lobbying στην Επιτροπή Ήτρε ή οποιαδήποτε άλλη. Γι' αυτό για μένα η Επιτροπή σας έχει τόσο σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας υποστηρίζει και να είμαι ξεκάθαρος για το τι μπορούμε να δεχτούμε και τι όχι όσον αφορά. Τώρα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πει στη διαδικασία επί παραβάση, υποθέτω ότι ενημερώνεστε. Θα το κοιτάξω πάντως, γιατί είναι η μία ή άλλη αναφορά η οποία οδηγεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε διαδικασία επί Αν τώρα υπάρχει ένα μοντέλο βάσει των οποίων φτάνουν οι αναφορές, Στη νέα συμφωνία με τα τρία θεσμικά όργανα για την καλύτερη νομοθέτηση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία. Είτε για την πλατφόρμα Refit, είτε για οτιδήποτε άλλο. Βλέπω δηλαδή να υπάρχει σύνδεση. Δεν είμαστε όμως μόνο εμείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μόνο του μπορεί να κοιτάξει ποιος είναι ο δικός του ο ρόλος απέναντι στα μέσα που διαθέτουμε. Για την ερμηνεία τώρα του άρθρου 51. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσω με την Επίτροπο Γιούροβα, κυρίως, για να δω πού βρισκόμαστε. Γιατί εσείς το έχετε θέσει ξανά και ξανά. Και θέλω να προσπαθήσω να δω από κοντά πόσο περιοριστική είναι η ερμηνεία του άρθρου αυτού και τι μπορούμε να κάνουμε. Η Επίτροπος Γιούροβα είναι αρμόδια και θέλει πολύ να το προχωρήσει. Θα πρέπει να μιλήσω μαζί της. Θα το κάνω. Για το Μαρακές, φυσικά και η Επιτροπή θέλει να εφαρμοστεί η συνθήκη γρήγορα υποβάλαμε πρόταση στο Συμβούλιο προς κύρωση. Έχει μπλοκαριστεί τώρα στο Συμβούλιο εξαιτίας ε, της φύσης των ε, εξωτερικών αρμοδιοτήτων, κάτι που μας έρχεται συχνά. Ζητήσαμε ε, γνώμη του δικαστηρίου, προδικαστική, και περιμένουμε τώρα τι θα μας πει και από εκεί και πέρα ελπίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να κυρωθεί η συμφωνία ετοιμάζουμε και το σχέδιο νομοθεσίας έτσι ώστε να ενταχθεί στο κοινοτικό δίκαιο άπαξ και πάψει το μπλοκάρισμα αυτό. Και έγκαιρα θα σας ενημερώσουμε τώρα. Οι ανταλλαγές πληροφοριών. Η κατάσταση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη έδειξε ότι το γεγονός ότι δεν ανταλλάζουν οι μυστικές υπηρεσίες τα δεδομένα τους οδηγεί σε τεράστια προβλήματα και επιτρέπει τρομοκράτες να μετακινούνται χωρίς πρόβλημα. Όμως, αυτό που είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει μία τέτοια δομή και οι κατάλληλες νομικές εγγύσεις και νομικές και δημοκρατικές, τότε τα δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται καλύτερα. Καλύτερα από σε αυτή την πεσοβέζικη κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Ναι, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και δημοκρατικός έλεγχος, αλλά και νομικός έλεγχος, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι και νομικά και δημοκρατικά στέκουν αυτά που κάνουμε. Τώρα, Συμφωνώ μαζί σα ότι συχνά αργούν οι απαντήσεις μας. Περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και αυτό γιατί καθυστερούν οι χώρες μέλη. Σέρνονται. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία ενό επόμενου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και να θέσουμε το ζήτημα αυτό της καθυστέρησης των απαντήσεων ώστε να συμφωνήσουν και οι χώρες μέλη ότι θα απαντάνε πιο γρήγορα σε μας. Θα φροντίσω να το θέσω στο επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Θα το θέσουμε σε πολιτικό επίπεδο, γιατί πράγματι βλέπω και εγώ ότι αυτή η καθυστέρηση, επαναλαμβάνεται αυτό που είπε η κυρία Καμπεσόν, είναι σωστό. Απάντησα και για το τι είναι παραδεκτό και τι όχι, όσον αφορά. Για τα παιδιά τώρα. Θέλουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με τις χώρες μέλη. Δεν μπορούμε να τις υποχρεώσουμε. Επ' είχα μακρά συζήτηση με την Επίτροπο Γιούροβα σήμερα το πρωί. Γιατί θέλουμε να θέσουμε το θέμα της προστασίας των παιδιών για πολλούς λόγους. Θα έρθει με αυτό το ζήτημα στο Κοινοβούλιο. Όχι ειδικά Ανταλλαγέ πληροφοριών για περιπτώσεις υιοθεσία, αλλά γενικότερα. Με τη μεταναστευτική κρίση κυρίως βλέπουμε παιδιά, παιδιά και γυναίκες να υποφέρουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε να τους προστατεύουν περισσότερο οι εθνικέ αρχές. Όπου μπορούμε λοιπόν θα το φροντίσουμε. Με ανησυχεί ιδιαίτερη κατάσταση. και γιατί οι ασυνόδευτοι, οι ανήλικοι φτάνουν στην Ευρώπη και ποιος ξέρει τι τύχη τους επιφυλάσσεται, αλλά και το θέμα της επανένωσης οικογενειών με προβληματίζει. Μερικές φορές είναι δύσκολο. Και τα παιδιά είναι αυτά που υποφέρουν περισσότερο. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ώστε οι χώρες μέλη να κάνουν το σωστό. Το θέμα τώρα της σύγκρουσης συμφερόντων. Όπως είπα, ας αρχίσουμε με περισσότερη διαφάνεια σε όλα τα θεσμικά όργανα. Σίγουρα εσείς θα με υποστηρίξετε πάρα πολύ σε αυτό. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχετε και τη δικιά σας δουλειά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το πω ομά, γιατί ούτε και εδώ τα πράγματα είναι τέλεια όσον αφορά τη διαφάνεια. Τώρα, η διαφάνεια βέβαια δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την διευκρίνηση των θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων. Αλλά είναι κοντά αυτά τα δύο. Για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τι πρωτοβουλία θα πάρουμε. Ελπίζω μέχρι τα τέλη της χρονιάς να έχουμε υποβάλει μια τέτοια πρωτοβουλία πριν τα τέλη της χρονιάς. Για την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών Ξέρετε ότι εξετάζουμε την αναθεώρηση του μέσου αυτού. Είναι πολύτιμο και γι' αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Το έχουμε ήδη συζητήσει αρκετές φορές με το Κοινοβούλιο. Και εγώ έχω δεσμευτεί να φροντίσω να γίνει ακόμα μεγαλύτερη η επιτυχία αυτό το μέσο. Όμως τα ζητήματα παραμένουν. Υπάρχουν περιορισμοί στην ίδια τη συνθήκη για το πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο. Σέβομαι απόλυτα τους πολίτες οι οποίοι λένε ναι, ωραία, συμφωνία, αλλά εμείς εδώ ανησυχούμε και θέλουμε να λάβουμε μια πρωτοβουλία ως πολίτες. Ναι, αλλά ως θεματοφύλακας των συνδικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια που τις θέτει η ίδια η συνθήκη. Βέβαια, ίσως να μπορέσει να υπάρξει με ρύθμιση κάποια βελτίωση στα ζητήματα εκείνα τα οποία κρίνονται προβληματικά για τους πολίτες. Αυτά προς το παρόν. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε με τους ομιλητές τώρα. Όλοι θέλουν να πάρουν τον λόγο. Ο κύριος Μαριάς τώρα, εκ μέρους του ECR. Και μετά ο κύριος Κύρκος. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας θα σας θέσω αυτό το θέμα που έχω θέσει ορισμένες φορές στην Ολομέλεια όταν συζητούμε, αλλά εκεί δεν έχουμε την άνεση να γίνει ένας διάλογος. Το θέμα αφορά το ρόλο της Κομισιόν στο πλαίσιο της Τρόικας, διότι συμμετέχει ως μέλος της Τρόικας και φυσικά διαπραγματεύεται με την ελληνική κυβέρνηση. Και υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες καταλήγουν εν συνεχεία με τη μορφή ενός μνημονίου συνεννόησης, Memorandum of Understanding. Πολλές φορές έχουμε θέσει το θέμα ότι το μνημόνιο συνεργασίας παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία υπάρχουν ε, και τα οποία υπάρχουν και προστατεύονται από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είχε τεθεί μια ερώτηση στην Κομισιόν η οποία πίντησε ότι, και θα σας το διαβάσω αγγλικά,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 επειδή ακόμα και αν η ΙΟΝΕ δεν είναι ευρωπαϊκή πράξη, αλλά είναι πράξη ανάμεσα στην Ελλάδα και την, τους δανειστές είναι εκτός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης. που έχει δώσει η Κομισιόν. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, διότι το μνημόνιο συνεννόησης εμπεριέχεται εν συνεχεία στις αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ και το ΕΚΟΦΗΝ εκδίδει μια απόφαση η οποία είναι δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως εδώ πρέπει λίγο να δείτε το θέμα της λειτουργίας της Κομισιόν. Συμμετέχει στη διαπραγμάτευση, συμφωνεί ένα Memorandum of Understanding και εν συνεχεία το ίδιο το ΕΚΟΦΗΝ μετατρέπει το MOU σε απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ που σημαίνει ότι αυτό είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι EU law. Θέλω λοιπόν να δείτε το θέμα και ουσιαστικά και τυπικά. Αν δηλαδή μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του μνημονίου στην Ελλάδα να παίρνει αποφάσεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουμε τέτοιε αποφάσει, διότι μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται οι συντάξει που είναι περιουσιακό δικαίωμα, μειώνονται οι δαπάνε οι δημόσιε και έτσι δεν έχουμε πρόσβαση στην υγεία και σε φάρμακα. Επομένω, έχουμε περιπτώσει τέτοιε. Θέλω λοιπόν να δείτε το θέμα αυτό ουσιαστικά. Πώ δηλαδή και ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να μην έχουμε παραβιάσει του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω του Μνημονίου Συνεννόηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο λόγος είναι για τον κύριο Κύρκο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ τον κύριο Τίμερμαντς και ειδικά επειδή είναι και υπεύθυνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα καταλάβει πιο καλά αυτά που θα του πω. Ε, στην Ελλάδα έχουμε προβλήματα με τη διαχείριση αποβλήτων, με τις παράμονομες χωματερές, με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από το 88 που είχε γίνει η πρώτη καταγγελία μέχρι σήμερα έχουμε καταλήξει μετά από διαδοχικές οι αποφάσεις δικαστηρίου να πληρώνουμε 20.000 ευρώ τη μέρα για τις χωματερές μας. Είναι μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται, όπως είπε και ο συνάδελφος, σε ε, μνημόνιο. Ε, πριν από λίγες, λίγους μήνες ε, φτιάξαμε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που ακολουθήθηκε με ένα στρατηγικό σχέδιο πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. Από νόμους είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια σχέδια είχαμε. Μέχρι το 2020 θα υπάρχουν 2,5 δισεκατομμύρια για την προστασία του περιβάλλοντος και 1 δισεκατομμύριο ειδικά για την διαχείριση των αποβλήτων. Πώς όμως μπορεί η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι αυτή τη φορά έστω, όχι όπως τις προηγούμενες, αυτά τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Δεν θα προσθεθούν σε έργα τα οποία είτε είναι άχρηστα, είτε δεν είναι λειτουργικά, είτε είναι λίγα, ώστε να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί σας λέω, από το 88 δεχόμαστε καταγγελίες εδώ για το περιβάλλον και έχουμε καταλήξει να πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα και η Κομισιόν συνεχίζει και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δίνει χρήματα για αυτό το ζήτημα και αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Τι μηχανισμούς ελέγχου έχετε τελικά ώστε να μην φτιάχνουμε σχέδια αλλά δεν, υλοποιούμε, δεν τα υλοποιούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. And now the floor goes to Paul from the e Ο λόγος από το ΑΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Τιμερμάνη, αναφέρατε την ε, πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών πριν από λίγα λεπτά και έχω μία ερώτηση για σας. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρεί ε, πολύ νωρίς να αρχίσει η διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας και από την άλλη υπάρχουν και οι προτάσεις του Κοινοβουλίου για την βελτίωση οι οποίες δεν εισακούονται. Θα μπορούσατε να μας πείτε στην πράξη πώς προτείνεται να βελτιωθεί η διαδικασία αυτή χωρίς να τροποποιηθεί η νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνεργασία του Κοινοβουλίου μας με εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία που έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου, δεν ακούγεται. Έχω διάφορες ερωτήσεις για σας. Αλλά μια από τις απαντήσεις που δώσατε στον προηγούμενο γύρο με εξέπληξε, οπότε αφήνω τις ερωτήσεις μου στην πάντα και θα επικεντρωθώ μόνο σε αυτή την καινούργια μου ερώτηση. Λέτε ότι για σας κάνει διαφορά το αν πρόκειται για ατομικές αναφορές ή αν πρόκειται για συλλογικές αναφορές ανθρώπων που είναι οργανωμένοι με μια εκστρατεία από πίσω τους, αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε. Με εκπλήσει λοιπόν αυτό, γιατί βλέπω να επαναλαμβάνονται ζητήματα. Για τα ζώα, για παράδειγμα. Πάρα πολλές αναφορές που μας στάνουν έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των ζώων. Η μεταφορά των ζώων, δοκιμές, πειράματα που γίνονται στα ζώα, πώς θα ανατώνονται στην Ισπανία, στη Ρουμανία. Θέματα τα οποία γνωρίζουν οι συνάδελφοι βέβαια πολύ καλά εδώ. Σήμερα το πρωί είχαμε μια οργάνωση που έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές σχετικά με την μεταφορά των ζώντων ζών. Συγκέντρωσε η οργάνωση λοιπόν όλες αυτές τις ε, υπογραφές και ήταν εδώ σε δάκρυα η κυρία που εκπροσώπησε την ε, οργάνωση αυτή που έχει υποβάλει την αναφορά επειδή λέει ήταν η πρώτη φορά που άκουσε καλά λόγια ενώ και δεκαετίες τώρα αγωνίζεται για την ευζοία λέει ότι η Επιτροπή ποτέ δεν τους αντιμετωπίζει με καλοσύνη. Πρώτη φορά ένιωσε υποστήριξη και εμένα αυτό με άγγιξε πραγματικά. Οπότε δεν βλέπω γιατί την υπάρχει αυτή η διαφορά. Και με εκπλήσει που αφήνουμε τον κόσμο να περιμένει και δεν εξυπηρετείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικές φορές το έχει πει και ο διαμεσολαβητής ότι εσείς σαν θεματοφύλακας των συνθήκων ε, πρέπει να συμπεριφέρεστε με περισσότερη, πώς να το πω, να συμπάσχετε περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να αντιμετωπίσετε σοβαρά και τέτοιε αναφορέ που δεν είναι ατομικέ αλλά που έχουν την υπογραφή πάνω από ένα εκατομμύριο ατόμων. Ευχαριστούμε. Μπέκερ, τελευταίος ομιλητή. Εκτό μικροφώνου, δεν ακούγεται το μικροφώνο του. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών και να διατυπώσω κάποιες σκέψεις που έχω. Η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί απαρτία ενός εκατομμυρίου πολιτών από ε, κάθε κράτος ε, μέλος και αυτό δεν γίνεται πρακτικά. Οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτών, αν το εξετάσουμε, είναι η εξής μία. Η πρωτοβουλία για το νερό. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι δεν επιθυμώ να ζω σε, ε, καμία χώρα που δεν έχει συνδικάτα και που δεν έχει ε, σωστή ε, οργάνωση, σωστή κοινωνική πρόνοια. Μία πρωτοβουλία λοιπόν Ευρωπαίων πολιτών είναι ένα μέσο το οποίο έχει δημιουργηθεί για, για την κοινωνία των πολιτών και όχι για τα, ε, τους κατεστημένους πολιτικούς θεσμούς οι οποίοι θέλουν να ρυθμίσουν, να ρεγουλάρουν αν θέλετε την πρόσβαση των ε, πολιτών. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία για το νερό είχε μία πολύ θεμητή βάση και ήταν επιτυχημένη μόνο επειδή τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ε, ασχολήθηκαν και έκαναν μία πολύ μεγάλη εκστρατεία. Ε, υπάρχει, υπήρξε λοιπόν κατάχρηση της πρωτοβουλίας των πολιτών. Από αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι υπάρχουν δύο ειδών καταχρήσης. Η μία είναι πολιτική και η άλλη είναι ηθική. Γίνεται κατάχρηση ενός μέσου το οποίο έχει δημιουργηθεί για τελείο σε διαφορετικό σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Πιτέρα. Δεν έχω ξεχάσει κάποιον άλλον. Κυρία Πιτέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Αντιπρόεδρο. Στις αναφορές που εξετάζουμε στην Επιτροπή μας, πολλές φορές είχαμε αναφορές για την απασχόληση και θυμάμαι δύο ιδιαίτερα από την Πολωνία οι οποίες είχαν εστιάσει στο εξή θέμα. Στην υπογραφή συμβάσεων εργασίας κενών. Εγώ αυτό το ονομάζω σύγχρονη δουλεία. Άνθρωποι που δεν έχουν παιδεία ε, ζητήθηκε να υπογράψουν άδεια σύμβαση εργασίας χωρίς ε, να ξέρουν τους όρους και πολλές φορές ε, το έχω φέρει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ρώτησα να μάθω εάν υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών και η απάντηση ήταν θετική και ξέρω πως υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις και σε άλλα κρατημέλη. Και ξέρω επίση ότι τουλάχιστον 12 κράτη-μέλη, ε, τα περισσότερα από αυτά νεότερα κράτη-μέλη, ε, τέθησαν υπό έρευνα για αυτό. Και θυμάμαι πως είχαμε και έναν νομικό εκπρόσωπο από το τμήμα ανάλυσης που μας εξήγησε ακριβώς γιατί έχουν σημειωθεί παραβάσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που ε, αντί να έχουμε κάποια ανταπόκριση δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολλοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν είναι μορφωμένοι, δεν σκέφτονται παγκόσμια, σκέφτονται τις δικές τους ζωές. Εάν λοιπόν μπορούμε να δείξουμε στους απλούς αυτούς πολίτες ότι δουλεύουμε για εκείνου, τότε θα ήταν η καλύτερη λύση και όχι η υπερβολική γραφειοκρατία και η υπερβολική ε, διοίκηση. Να τους δείξουμε ότι υπάρχει κάποιος που υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό και θα ήθελα να κάνω έκκληση σε εσάς για ε, να λύσετε αυτό το πρόβλημα, να υπάρξει κάποιο σχέδιο, κάποια πρόταση. διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερε κλίμακα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα σας δώσω τώρα το λόγο, κύριε Τίμερμανς, να ολοκληρώσετε. Παρακαλώ, πάρτε το χρόνο σας και σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς και εγώ είχαμε ε, και στο παρελθόν ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά σήμερα. Και πολλές φορές δυσκολεύομαι να δω τη σχέση αυτών που λέει με την Επιτροπή Αναφορών. Ωστόσο γνωρίζω ότι ε, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον και τον σέβομαι πάρα πολύ διότι είναι δεσμευμένος ε, για αυτό το θέμα. Είναι πάντα παρόν σε κάθε ανταλλαγή απόψεων και ε, προσπαθεί να τοποθετηθεί πάντα. Γι' αυτό λοιπόν τον θαυμάζω. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να του δώσω την ίδια απάντηση που του δίνω κάθε φορά η οποία είναι ότι το πρόγραμμα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο ε, το πρόγραμμα της Τρόικα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και από τις ελληνικές αρχές. Έχουν περάσει επίσης εκλογές γι' αυτό το πρόγραμμα. αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε το πρόβλημα της ε, ανόδου του εξτρεμισμού στην Ευρώπη εάν η οικονομική κρίση δεν είχε τόσο ε, μεγάλες επιπτώσεις σε εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους και βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση που δεν αντέχουν οικονομικά να πληρώσουν ιατροφαρμακευτική υπερίθαλψη που δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο. Αφήνοντας λοιπόν κατά μέρο ε, την επίσημη θέση μου, την οποία έχω επαναλάβει στο παρελθόν, έχει επαναλάβει και ο κύριος Μαριάς, μένει μια πρόκληση, πρόκληση που για μένα αφορά θεμελιώδεις αξίες. Δεν αφορά κατά ανάγκη τα μεμονωμένα μέτρα που έχουν ληφθεί από μεμονωμένες κυβερνήσεις και έχουν πλήξει αυτές τις θεμελιώδεις αξίες, αλλά βλέπουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης να αμφισβητούνται οι θεμελιώδεις αξίες από πολιτικό εξτρεμισμό, από ξενοφοβία ε, κτλ. Υπάρχει σίγουρα σχέση ανάμεσα στην οικονομική κρίση και στην κρίση αξιών των πολιτών. Αυτό το βλέπουμε και με τη μεταναστευτική κρίση. Εάν καταφέρουμε, όχι να επιλύσουμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να λύσει αυτήν την τεράστια πρόκληση ε, που θα παραμείνει για τις επόμενες γενιές εδώ, εάν καταφέρουμε να την διαχειριστούμε έστω, να την ελέγξουμε, εάν μάλλον δεν καταφέρουμε να την ε, διαχειριστούμε, τότε θα αποχωρήσουν οι πολίτες από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποχωρήσουν από απελπισία και θα επαναλάβω ότι δεν συμφωνούμε ε, ως προς τις ε, ε, τελικές μας θέσεις, όμως σίγουρα αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της. Σε σχέση τώρα με τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα. Νομίζω πως με την πάροδο των ετών, των δεκαετιών, έχουμε καταλάβει πως πρέπει να είμαστε ε, πιο επαγγελματικοί στη δράση μας. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω κάποια επιστημονικά στοιχεία, αλλά θα πω ότι εάν τα κονδύλια που είχαν ε, προοριστεί για ε, την λύση του, του προβλήματος των ε, χωματερών στην Ελλάδα είχαν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό, τότε τώρα δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά βλέπω τρομερή βελτίωση και το λέω εγώ που είμαι και παλιά καραβάνα. Βλέπω τρομερή βελτίωση παρά τις τρομερά αντίξωες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να οικοδομήσουμε ε, το μέλλον. Τώρα, ε, σε σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου. Είμαστε πολύ κοντά στη θέση του Κοινοβουλίου. Αυτό το έχω πει και στο παρελθόν και θέλω να υπάρξει επιτυχής λύση όσο και εσείς. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να αλλάξουμε τον κανονισμό, όμως δεν θα έλεγα ότι το έχουμε αποκλείσει. Δεν έχουμε αποκλείσει να τροποποιήσουμε τον κανονισμό, πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και έχουμε απειροελάχιστες δυνατότητες να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θα καταφέρω να το κάνω. Διότι μην ξεχνάτε πως υπάρχει και το Συμβούλιο. Μπορεί εμείς να συμφωνούμε, η Κομισιόν και Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει και το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το... Ε, αυτή η προσπάθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο μέλλον για την βελτίωση της ε, συνεργασίας μας. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όχι ως τελευταία λύση επειδή δεν καταφέραμε να περάσουμε την νομοθεσία μέσω ε, των ε, συνηθισμένων διάβλων, αλλά και επικοδομητικά. Τώρα, με εκπλήσουν τα σχόλια της κυρίας Χάζεκαμπ διότι για όσους δεν γνωρίζετε η κυρία Χάζεκαμπ εκπροσωπεί ένα κόμμα το οποίο εναντιώνεται σε οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία. Ε, καταπολέμησε την ε, συνταγματική συνθήκη θερμότατα διότι δεν τους ευχαριστούσα ε, σε τα όσα προέβλεπε για τα δικαιώματα των ζώων. Δεν λάβαμε βέβαια κάποια αντιπρόταση παρά την άρνησή του στην συνταγματική συνθήκη. Και τίθενται επίσης την ε, Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία εξαιτίας της κατάστασης με τα πουλερικά εκεί. Και πάλι, ε, δεν έλαβα καμία απάντηση στην ε, ερώτηση του «Ωραία, απορρίπτουμε τη συμφωνία. Πώς αυτό θα βελτιώσει τη ζωή στα κοτόπουλα εκεί». Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως μπορώ να τονίσω αυτές τις ασυνέπειες ε, στις ε, απόψεις της. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι επιτρέπεται να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, όταν μας λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες, δεν μπορείτε να μας ζητάτε να αναλάβουμε και άλλες. Και πρέπει να αντιδράσω σε αυτό που είπατε, όπως και πρέπει να αντιδράσω και σε αυτό που είπατε για τα δικαιώματα των ζώων. Εδώ να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών έχουν πολύ ισχυρή άποψη για τα δικαιώματα των ζώων. Και εγώ επίσης πιστεύω ότι αν βελτιώσουμε την ε, διαβίωση και τα δικαιώματα των ζώων στην Ευρώπη, και ε, η κοινωνία μας και η οικονομία μας θα ε, βελτιωθεί και χρειάζεται σωστή ενημέρωση έτσι ώστε να προχωρήσουμε προς αυτή τη βελτίωση και είμαι σίγουρος ότι με τη σωστή ενημέρωση θα έχουμε την στήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών διότι θα μεγαλώσουν Ευρωπαίοι πολίτες σε μια κοινωνία όπου τα ζώα δεν θα είναι αντικείμενα αλλά θα έχουν καλύτερη μεταχείριση αντέδρασα στα θέματα που θίξατε πολιτικά, όμως ε, να είστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε αναφορά που σχετίζεται με τα δικαιώματα των ζώων θα έχει ε, την προσοχή που της αξίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες όταν γίνονται με το σωστό τρόπο θα έχουν την ε, δέουσα Προσοχή, η συνεισφορά των πολιτών είναι πολύτιμη και κάθε συνεισφορά, ακόμα και η μικρότερη, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά όταν συμμετέχετε σε ένα κίνημα πολιτών το οποίο μπορεί να οργανωθεί, όταν ως πολίτης κάνετε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή πιστεύετε ότι κινδυνεύουν τα δικαιώματά σας, η απήχηση θα είναι μεγαλύτερη εάν γίνεται από πολλούς μια πρωτοβουλία και όχι από ένα μεμονωμένο πολίτη. Το δικαίωμα στην αναφορά είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και ο σκοπός ήταν αυτός, ο, ο πολίτης δηλαδή, ο μεμονωμένος πολίτης να έχει πρόσβαση στην εξουσία. Και μέχρι τώρα έχουμε δει ότι τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά. Ε, και τέλος, όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας. Να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε δεσμευμένοι ο κάθε πολίτης να λαμβάνει ίσες ε, αποδοχές για ίση εργασία. Η σύγχρονη δουλεία είναι απαράδεκτη και το να εκμεταλλεύεται κάποιος την ε, αδύναμη θέση ενός ε, ανθρώπου στην αγορά εργασίας είναι απαράδεκτο. Κυρία Πιτέρα, θα κοιτάξω το θέμα προσωπικά, αλλά σίγουρα είναι λάθος να δημιουργούνται στην εποχή μας συμβάσεις εργασίας μηδενικών ορών συνθήκες μοντέρνας δουλείας Ίσως αυτό δεν ε, πρέπει να αφορά μόνο την Επιτροπή Αναφορών, αλλά είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τους ευάλωτους ε, πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε και θα χαρώ πολύ να συνεχίσω το διάλογό μας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ήταν προνόμιό μα να σας έχουμε σήμερα εδώ για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όχι μόνο εσάς προσωπικά, αλλά και το επιτελείο σας. Και να σας κάνω μια ξεκαθαρή δήλωση εκ μέρου τη επιτροπή μας, ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η συνεργασία μα και είναι πάντα χαρά μας όταν συνεργαζόμαστε με προσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αυτό θα το κάνουμε μαζί, όμως έχουμε βάλει τα θεμέλια και σίγουρα φέτος είναι καλύτερα από πέρυσι. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα και ανυπομονώ να συνεχίσουμε την καλή μας συνεργασία. Okay. So, this brings... Ωραία. Οπότε ερχόμαστε στο σημείο 23 της ημερησία διάταξης που είναι η αναφορά 2089 του Λουίτζι Τη Στέφανο σε σχέση με τη σύλληψη και κράτηση δύο Ιταλών αυτών στην Ινδία. Ο αναφέρον είναι εδώ και σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Buonasera. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους για την ευκαιρία που μου δίνετε. Έχω υποβάλει μια αναφορά σε σχέση με την υπόθεση των δύο δύο δύο Ιταλών πεζοναυτών που κρατούνται στην Ινδία εδώ και τέσσερα χρόνια. Είμαι ε, ειδικό ε, δικαστική ανάλυσης με 20 χρόνια εμπειρία πίσω μου και ήθελα να δείξω στην Επιτροπή σας ε, νέα στοιχεία που έχουν υπάρξει σε αυτή την υπόθεση από τότε που τον Αύγουστο του 2015 δημοσιεύθηκαν από το δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας του Αμβούργου τα Ινδικά δικαστικά έγγραφα τα οποία ε, κρατούν το απόρριτα από τις Ινδικές Αρχές εδώ και τέσσερα χρόνια. Το δικαστήριο λοιπόν μου τα παραχώρησε χωρίς ε, δέσμευση περί της χρήσης τους μετά από απλό αίτημα και από αυτά τα έγγραφα προκύπτει λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για τα ινδικά δικαστικά έγγραφα, προκύπτει λοιπόν από αυτά ότι οι δύο αυτοί πεζοναύτες είναι αθώοι και αυτό που είναι ακόμη πιο σοβαρό είναι ότι η αθότητά τους ήταν εν γνώση των Ινδικών αρχών τουλάχιστον από τη δεύτερη μέρα κράτησης, μάλλον δεύτερη μέρα μετά τα γεγονότα, όταν δηλαδή έγιναν οι αυτοψίες. Θα σας αναφέρω σύντομα ποια είναι τα έγγραφα. Εδώ βλέπετε την εμπειρία μου, το βιογραφικό μου. Η εμπειρία μου προέρχεται από τη συμμετοχή μου σε εξαιρετικά περίπλοκες υποθέσεις, πάντοτε στον τομέα της αεροναυπηγικής, τόσο στην Ιταλική εισαγγελία, όσο και σε ιδιωτικές υποθέσεις. Τώρα, εδώ, σύντομα λοιπόν θα σας παρουσιάσω όλα όσα μπορείτε να δείτε πιο εμπεριστατωμένα στο ειδικό site internet που έχουμε φτιάξει στα αγγλικά και που είναι ε, προσβάσιμο για όλους. Από την ημέρα των γεγονότων οι Ινδικές Αρχές γνωρίζουν ότι ανάμεσα στο περιστατικό του Ρίκα Λέξη του Ιταλικού δηλαδή πλοίου το οποίο κατηγορείται ότι ε, ε, παρέ, ότι πετέθησε Ινδικό αλληλευτικό σκάφος έχουν περάσει πέντε ώρες διαφορές. Από τη στιγμή της εισόδου στο λιμάνι, ο, ο, καπετάνιος του αλληλευτικού λέει ότι οι πυροβολισμοί ε, ακούστηκαν στις 21 και 30 και όχι στις 10. 7 και 30. Από το επόμενο πρωινό στο λιμάνι Κώση έρχεται ε, το ψευδές αλληλευτικό σκάφος Σαντ Το πραγματικό είναι σε 200 χιλιόμετρα στο ε, νότια, νοτιότερα, στο αλληλευτικό λιμάνι ε, που λέγεται Δεκάρα και αυτά όλα εν γνώση των ειδικών αρχών. Το απόγευμα της επόμενης ημέρα, 16 του μηνός, έγινε η αυτοψία. Η αυτοψία είναι διαθέσιμη μέσω του ε, δικαστηρίου για το δίκαιο της θάλασσας του Αμβούργου. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα βλήματα που βρέθηκαν στα σώματα των δύο θυμάτων δεν χρησιμοποιούνται από τους ιταλού από το Ιταλούς Αυτό αγνοείται και προχωρούν από την επόμενη μέρα στην σύλληψη των δύο πεζοναυτών. Οι αλληλείς στις 17, δηλαδή δύο μέρες μετά από τα γεγονότα, επιβάλλουν την πρώτη εκδοχή. Δηλαδή ότι οι πυροβολισμοί και αυτό σε, σε, σε δημόσια συνέντευξη βλέπετε στην εικόνα του αλληλείς που περιγράφουν τι έγινε. Λοιπόν, στις 17 του μηνός επιβεβαιώνουν ότι οι πυροβολισμοί έγιναν βράδυ, ενώ εκείνοι βρίσκονταν στα είδατα της Ινδίας, δηλαδή στα 12 μίλια από την ακτή και όχι στα 20 μίλια, όπως, όπου αντίθετα βρισκόταν το Ιταλικό σκάφος. Κάλλη μια απόδειξη την οποία γνώρισε το Ινδικό δικαστήριο ότι η δική μας είναι αθώοι. Επι... Τώρα, επιπλέον, η επιτόπου έρευνα που έγινε από τις συνδικές ε, αρχές μετρά της ενώ μετράμε με ζούρα, μετρά την διάμετρο των Ιταλικών βλημάτων ε, μέχρι τελευταίο χιλιοστού. Και με βάση αυτή την αυτοψία που καταλήγει ότι είναι 55-56, δηλαδή εκατοστά χιλιοστού, ε, με βάση αυτή την αυτοψία συλλαμβάνονται οι στρατιώτες μας. Παράβαση του δικαιώματος αμήνης στις 29 Φεβρουαρίου του 2012, το δικαστήριο του Κόλαμε αρνείται στους Ιταλούς εμπειρογνώμων να συμμετέχουν στην ε, βαλιστική επαλήθευση η οποία θα γίνει τη απουσία των ε, υπερασπιστών των ε, κατηγορουμένων. Σε οποιοδήποτε δικαστήριο δεν ισχύει τέτοια διαδικασία και άρα ολόκληρη διαδικασία θεωρείται άκυρη. Η βαλιστική έρευνα ε, των ειδικών αρχών παρουσιάζεται ως απόδειξη της ενοχής των Ιταλών πεζών αυτών. Αλλά γιατί, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει, αρκεί να τη διαβάσουμε, ε, καθίσταται απόρριτη. Οπότε, Βλέπουμε σε αυτή την αυτοψία ότι τα βλήματα που βρέθηκαν στα σώματα των δύο θυμάτων είναι περίπου παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιεί το Ιταλικό, το Ιταλικό στρατός. Περίπου. Αυτό αποδεικνύει την αθωότητα των δύο στρατιωτικών μας. Ένα ακόμα σημείο σημαντικό για την Ινδική βαλιστική έρευνα είναι ότι υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στο, σε ένα κομμάτι βλήματος και το, τα όπλα των πεζοναυτών. Αν γίνει ανάλυση τρισδιάστατα, επαληθεύουμε ότι εδώ πρόκειται για ακόμα μια απόδειξη της αθωότητας των Ιταλών πεζοναυτών, διότι αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να προέρχεται από όπλο ε, διαμέτρου 56 χιλιοστών. Τώρα, το αλευτικό σκάφος Αντάντονη, αφού αναλύθηκε από τους Ινδούς ανακριτές, επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη που το αφήνει να βυθιστεί. Δηλαδή δεν μπορούμε η υπεράσπιση να επανέλθει και να κάνει αναλύσεις και έρευνες επί του αλλιευτικού αυτού σκάφους και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή δεν προστατεύτηκε ε, μία, ένα αποδεικτικό στοιχείο και αυτό οδηγεί στην ακύρωση κανονικά της δικαστικής διαδικασίας. Τώρα, στο παράτημα 48 και έχουμε και προσαρτημένο έγγραφο για ότι εδώ αυτό το έγγραφο υποβλήθηκε στο δικαστήριο του Αμβούργου και βλέπουμε το, τη σκηνή του εγκλήματος όπου το ιταλικό σκάφος ε, παρουσιάζεται ότι βρισκόταν σε λανθασμένη θέση κατά 20 μοίρες ενώ η θέση του ιταλικού σκάφους αναλύεται από ένα συναγερμό που χτύπησε γιατί η θέση του ήταν σωστή και άρα τα χτυπήματα θα είχαν, έρθει, θα είχαν χτυπήσει αριστερά το αλευτικό σκάφος, ενώ έτσι όπως υποτίθεται ότι βρισκόταν θα το είχαν χτυπήσει από τα δεξιά. Άρα λοιπόν υποβάλλεται ψευδές έγγραφο ώστε να επικυρωθεί η ενοχή των δύο παίζων αυτών. Παρακαλώ, μήπως μπορείτε να ολοκληρώσετε. Σας έδωσα πέντε λεπτά, ήδη ξεπεράσατε κατά δύο λεπτά το χρόνο σας. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν να ολοκληρώσετε και θα έχετε το λόγο μετά από τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήδη καταλάβαμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Σας ευχαριστώ. Τον Ιανουάριο του 2015 το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε ψήφισμα όπου στα δύο του σημεία Α και Β θεωρεί βέβαιο ότι οι Ιταλοί πεζοναύτες πυροβόλησαν εναντίον του αλευτικού σκάφου Αντάντονη. Αυτό δεν είναι αλήθεια και κανένα ειδικό ε, ε, έγγραφο δεν το αποδεικνύει αυτό. Βασίζονται μόνο σε συγκυρίες, σε μαρτυρίες οι οποίες έχουν αυτοδιαψευστεί διότι ο καπετάνιος του αλλιευτικού θα αλλάξει μετά εκδοχή και θα πει ότι ε, το περιστατικό συνέβη στις 4.30. Άρα λοιπόν το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παραπλανήθηκε από παραπληροφόρηση την οποία διέδωσε οι αρχές της Κεράλα. και καλή την πίστη αυτέ οι αποδείξει υποβλήθηκαν στο δικαστήριο του Αμβούργου για το δίκαιο τη θάλασσα. Άρα λοιπόν αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διορθωθεί. Εγώ ζητώ να οριστούν τέσσερι εμπειρογνώμονε, όχι Ιταλοί, από την Επιτροπή σας που θα ζητήσουν από το Δικαστήριο του Αμβούργου τα ίδια τα, αυτά, τα ειδικά έγγραφα που εγώ έλαβα και που θα επαληθεύσουν τα όσα εγώ υποστηρίζω. Εάν λοιπόν εσείς ορίσετε τέσσερις επιγνώμονες και σε περίπτωση που θελήσουν να με δικαιώσουν, τότε αυτό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να διορθωθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα δίνω το λόγο στους ε, στην εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση που μπορεί να μας δώσει κάποια παραπάνω στοιχεία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Από το Φεβρουάριο του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την περίπτωση αυτή των δύο Ιταλών πεζοναυτών μαζί με την Ιταλική κυβέρνηση. Η κατάσταση συνεχίζεται τέσσερα χρόνια τώρα, όπως είπε ο αναφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ζήτησε επανειλημμένως μια γρήγορη λύση προς το συμφέρον και της Ιταλίας και της Ινδίας βάσει του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα της σύμβασης για την θάλασσα του ΟΗΕ. Τώρα έχει υποβληθεί η περίπτωση σε διεθνή διαιτησία και τόσο η Ινδία όσο και η Ιταλία έχουν δεσμευτεί στην διαδικασία αυτή διαιτησίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αναφερθεί σίγουρα θα υπάρξει απόφαση μετά τις ακροάσεις που έλαβαν χώρα 30 και 31 Μαρτίου. Η διάσκεψη κορυφής που έλαβε χώρα στις 30 Μαρτίου Ινδίας Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έδωσε την δυνατότητα να επαναλάβουμε τις ανησυχίες μας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είπε στην Ινδία επί ευκαιρία της διάσκεψης αυτής ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες της Ιταλίας όσον αφορά την κατάσταση των δύο αυτών Ιταλών αυτών. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα και από την Λία και από την Ινδία για να καταλήξει η περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Είναι πιο ξεκάθαρα τώρα τα πράγματα. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους συναδέρφους να κοιτάξουν και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου που λένε ξεκάθαρα ποια είναι η δικιά μας η θέση. Οι συνάδελφοι τώρα παρακαλώ. Δεν έχεις δίσει κανείς το λόγο μέχρι τώρα. Και ξαφνικά έγινε η Ιταλική η αίθουσα εδώ. Όλοι σχεδόν οι ευρωβουλευτές παρόντες είναι Ιταλοί. Οι Πολωνοί και οι Σουηδοί είμαστε μειονότητα εδώ. Ο κύριος Μπορκέζη έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω ως Ιταλός πολίτης αλλά και ως Ευρωπαίος πολίτης για την προσοχή που έχει δώσει αυτή η Επιτροπή σε μια υπόθεση εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο όπως μπορεί να φανεί ε, λόγω της παρουσίας τόσων ε, Ιταλών Ευρωβουλευτών, γιατί πρόκειται για ειδικά Ιταλικό ενδιαφέρον, αλλά για ευρωπαϊκό, και για ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, γιατί εγώ εδώ Βλέπω πολύ σημαντικό, δεν βλέπω μάλλον τις λεπτομέρειες τις τεχνικές, γιατί δεν έχω τις ε, ακατάλληλες γνώσεις. όλοι έχουμε εκτιμήσει τον χαρακτήρα σοβαρό της ε, υπόθεσης υψηλού επιστημονικού επίπεδου που μας εξέθεσε ο κύριος ε, Ντιστέφανο. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω για μια άλλη άποψη. Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Θα πρέπει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που ξέρω ότι μελετά αυτό το θέμα να επιμείνει περισσότερο ή ε, να παρέμβει πιο έντονα. Γιατί θα πρέπει εδώ να φωτιστεί αυτή η τόσο σημαντική πτυχή. Αυτοί οι πολίτες μας βοηθήθηκαν πολύ ε, αδύναμα επιτρέψατε μου να πω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ αυτό το πρόβλημα θέλω να αναφέρω. Θεωρώ ότι κάθε λάθος μπορεί να διορθωθεί και ίσως ε, σήμερα θα πρέπει να αλλάξουμε ε, στάση. Από τα όσα μας παρουσιάστηκαν δεν νομίζω και ότι υπάρχουν αντίθετα στοιχεία από το όσα μας είπε αναφέροντας. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, τα ενδικά, προκύπτει προφανώς πόσο έγιναν προσπάθειες ε, χειραγώγησης αυτών των στοιχείων και που προκάλεσαν μια βιαστική απόφαση, ειδικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα έπρεπε λοιπόν περισσότερο να πιέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να το αναλάβει και να πολύ αποφασιστικά και έντονα να παρέμβει, γιατί εδώ βρισκόμαστε πέρα από το ότι έχουμε φούμος πουρσεκουζιώνης, έχουμε και το αρρώστουμ περσεκουτσιόνους, δηλαδή δυο εργαζόμενοι Ευρωπαίοι που βρίσκονται σε αποστολή. Δεν έκαναν τουρισμό στην Ινδία. Πρέπει να υπερασπιστούμε τη, ε, ε, ε τους ανθρώπους ήταν εκεί για να δουλέψουν κατά της διεθνούς πειρατείας. Εμείς το στείλαμε για να υπερασπιστούν αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες. Αλλά εμείς μετά δεν τους υπερασπιστήκαμε όπως έπρεπε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Στάκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω στον Ιταλό φίλο μας ότι εγώ δεν είμαι Ιταλός, ανήκω στην Ουγγαρι... Ουγγρική μειονότητα της Σλοβακίας. Ακούτε τη διερμηνία, ρωτάει. Ναι. Θα αρχίσω από την αρχή. Πρέπει να πω λοιπόν ε, στους τέλους φίλου μου ότι δεν είμαι Ιταλός αλλά ανήκω στην Ουγγρική μειονότητα της Σλοβακίας. Ε, γιατί είπε η πρόεδρο πιο πριν ότι οι Σουηδοί και η Πολωνία Πολωνοί είναι μειονότητε σε αυτήν την αίθουσα. Όχι, όχι, είμαι κι εγώ. Το ΕΛΚ μου ζήτησε να τοποθετηθώ σε αυτήν την ε, αναφορά. Νομίζω πως εδώ έχουμε ένα θετικό βήμα. Το θέμα δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών της Ινδίας, έχει προχωρήσει βρίσκοντας στο Αμβούργο και πιστεύω πως η επιχειρηματολογία είναι μεν ε, πιστική, όμως η απόφαση δεν πρέπει να ληφθεί βιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε τι θα αποφασιστεί στο Αμβούργο. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες του θέματος και να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή, να μην αποφασίσουμε οριστικά σήμερα. Ο κύριος Καστάλντο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε σε σχέση με το όσα έλεγε ο συνάδελφος Σάκη προηγουμένως, είναι σωστό ότι δεν είναι μόνο αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής το να υποκαταστήσει την εργασία του δικαστήριο του Αμβούργου. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα στοιχεία που μας υπέβαλε ο αναφέρον σήμερα, διότι εάν επαληθευτούν όλα αυτά, πραγματικά θα σήμαιναν μια καταφανή παραβίαση των δικαιωμάτων που θα έπρεπε να είναι εγγυημένα για αυτούς τους ανθρώπους ε, και με το παραπάνω για ανθρώπους ε, οι οποίοι στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία και μάλιστα κατηγορήθηκαν αδίκως. Ε, είναι σαφές ότι σε αυτή την υπόθεση, εάν όντως επαληθευτούν όλα αυτά, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε γιατί θυμίζω ότι η Ινδία όπως είχαμε τη δυνατότητα να το θυμίσουμε και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, για το ψήφισμα το οποίο προναφέρθηκε, έχει συνυπογράψει και κυρώσει το σύμφωνο για τα ε, πολιτικά και αστικά δικαιώματα, διεθνή σύμβαση που εγγυάται μια ολόκληρη σειρά στάνταρ δικαιωμάτων για ένα σωρό και για όσους ε, υπόκεινται σε διαδικασία ποινική φύση. Ε, και αυτό το λέω για να επαναλάβω ότι σε αυτό το πλαίσιο οι δύο αυτοί πεζοναύτες είναι δύο πολίτες, όχι μόνο Ιταλοί, αλλά Ευρωπαίοι. Γι' αυτό και ζητάμε εντόνως την στήριξη από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την ΣΥΠΑ της εκπροσώπου. Γνωρίζουμε πως αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση η περίφημη ανανέωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με την Ινδία. Αν λοιπόν από πλευρά των Ινδικών Αρχών δεν επιδειχθεί διαφάνεια και τίμια διαδικασία χωρίς καμία μάλλον πλήρως αμερόληπτη πράγμα το οποίο όπως γνωρίζουμε δεν ε, τηρήθηκε ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσες ποιώσεις ασκήθηκαν σε αυτή την υπόθεση ώστε να ε, καταστεί πολιτική υπόθεση στις τελευταίες εκλογές ε, θέλουμε λοιπόν να αναλυφθούν μέτρα ως προς αυτή και περιμένοντας και σεβόμενοι βεβαίως την απόφαση του δικαστηρίου του Αμβούργου ζητάμε τη στιγμή που επιβεβαιωθούν αυτές οι ευθύνες να τεθεί επιτάπητος η μία ανανέωση αυτής της συμφωνίας και άλλα μέτρα ώστε να τιμωρηθεί η χώρα αυτή ε, επειδή ε, φυλάκισε δύο ανθρώπους χωρίς να ακολουθήσει μάλιστα την σωστή και διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κοτσολίνο. Και εγώ σύντομα εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την τεκμηρίωση που μας ε, παρουσιάστηκε σήμερα. Και μάλιστα επειδή είμαι και έχω παρακολουθήσει όλη αυτή την υπόθεση μέσω των πληροφοριών που <coughs> διαβάσαμε στις εφημερίδες. Γιατί είδαμε σιγά σιγά τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Πολύ εντυπωσιακά λοιπόν τα όσα μας αναφέρατε. Είναι προφανές ότι εμείς ε, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να παρέμβουμε εφόσον τρέχει η δικαστική διαδικασία. Διεθνή διατησία. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα όλη αυτή η διαδικασία και καταρχάς για το θέμα το πιο ουσιαστικό, δηλαδή την ε, περιορισμό της ελευθερίας των δύο παίζων αυτών. Είναι ακόμα στη φυλακή. Πέρα από την ουσία της συζήτησης, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και το θέμα της ελευθερίας ε, μετακίνησης είναι καθοριστικό, πέρα από τις κατηγορίες, τις αποφάσεις κτλ. Ίσως όμως θα πρέπει να αξιολογήσουμε και πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά, να μην κλείσει αυτή η συζήτηση, να επανέλθουμε δηλαδή μόλις θα υπάρχουν εξελίξεις. Ίσως μπορούμε να προωθήσουμε μια πρωτοβουλία σε επίπεδο του Κοινοβουλίου ως Επιτροπή Αναφορών. Αφού λάβαμε όλη αυτή την τεκμηρίωση, μπορούμε να στραφούμε στους συναδέλφους και ε, βουλευτές Ινδούς, ίσως μια πρωτοβουλία της Προέδρου προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν απαραίτητη από πολιτικές άποψεις. Δεν ε, παρεμβαίνει, δεν επηρεάζει την δικαστική διαδικασία για τη αλλά καλεί τους ε, συνάδελφους Ινδούς βουλευτές για αυτή την, σε μια, για αυτή την υπόθεση και αυτή την τεκμηρίωση που είναι πολύ καλά καλά παρουσιασμένη και που επιβεβαιώνει αυτό που ούτως ή άλλως εμείς στην Ιταλία ήμασταν σχεδόν βέβαιοι ότι ίσχυε, δηλαδή την αθωότητα των δύο όπεζων αυτών. Αυτή την πρόταση έχω να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, στρέφομαι στον κύριο Τη Στέφανο. Έχετε και πάλι το λόγο για τα συμπεράσματα. Δύο λεπτά το πολύ παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο ο Εντάξει τώρα, Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για τις παρεμβάσεις σας και για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε, ότι δηλαδή να δοθεί εκ νέου προσοχή σε αυτή την υπόθεση. Εγώ ως τεχνικός, διότι Εγώ έρθει εδώ ως τεχνικός, ως εμπειρογνώμονας ε, δικαστικής ανάλυσης. Ε, θέλω να επαναλάβω ότι από τη δεύτερη μέρα μετά τα γεγονότα οι ειδικέ αρχές γνώριζαν ότι οι δικοί μας ήταν αθώοι. Γιατί τα βλήματα που βρέθηκαν στα θύματα δεν περνάνε από τις σκάνες των όπλων τους γιατί είναι πολύ μεγάλες οι σφαίρες δεν μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί από αυτά τα όπλα και όλα αυτά κρύφτηκαν λόγω του απορρίτου των δικαστικών γράφων τα οποία δεν δόθηκαν στην υπεράσπιση ούτε και στην Ιταλική Εισαγγελία που επανειλημμένως τα ζήτησε μέσω ε, των διεθνών διάβλων. Από τη στιγμή που είχαμε τα έγγραφα στα χέρια μας και φυσικά τα διαβάσαμε ως εμπειρογνώμονες γιατί πρόκειται για τεχνικό δικαστική ανάλυση, δεν πρόκειται για τίποτα το εύκολο, Προκύπτει λοιπόν αυτό το οποίο σας ε, παρουσίασα. Εγώ λοιπόν ως τεχνικός θα εναποθέτω όλα αυτά τα στοιχεία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητώ δεν, σας, δεν απαιτώ να με πιστέψετε εμένα, αλλά μπορείτε να ζητήσετε αυτά τα δικαστικά έγγραφα που πλέον βρίσκονται στο, στο δικαστήριο του Αμβούργου και που είναι πλέον δημοσιευμένα, ε, γιατί όλα τα έγγραφα δημοσιεύονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, απόρριτα στοιχεία. Άρα λοιπόν να τα πάρετε κι εσείς αυτά τα έγγραφα και να είναι στη διάθεσή σας έτσι ώστε στις επαφές με την Ινδία, στις επαφές στις πολιτικές με τους Ινδούς βουλευτές να μπορείτε να συζητήσετε για την πραγματικότητα και, για όχι, και όχι για όλη αυτή τη σειρά των ψεμάτων που κυκλοφορούσαν εδώ και τέσσερα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να συνοψίσουμε τώρα. Τι έχουμε. Έχουμε δύο Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί σε μια τρίτη χώρα. Είναι, υποθέτω, νέοι. Δεν έχω λεπτομέρειες, αν έχουν συζύγους παιδιά, είναι Ευρωπαίοι πάντως. Και εδώ είμαστε για να προστατεύσουμε το μέλλον τους, την ευημερία τους και το παρόν τους βέβαια. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία διαιτησίας. Δεν μπορούμε να παρεύουμε σε αυτήν. Αυτό όμως που μπορούμε σίγουρα να κάνουμε είναι ότι θα κοιτάξουμε πάλι το ψήφισμα. Εγώ το έκανα. Μπορούμε να στραφούμε σε μία από τις αντιπροσωπείες του σώματος εδώ, τις αντιπροσωπείες δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις μας με την Ινδία και να ενημερώσουμε για την περίπτωση. Μπορούμε επίσης να στραφούμε προς τις αρχές της Ινδίας, την ε, αντιπροσωπεία δηλαδή των πρέσβη των Ινδό στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστολή μας, όπου να υπογραμμίζουμε τις δραστηριότητες της Επιτροπής μας επί του θέματος. Αυτό προτείνω λοιπόν να κάνουμε συνάδελφοι. Ξέρουμε ότι η διατησία λαμβάνει χώρα εκ παραλλήλου Οπότε εμείς, επειδή πρόκειται για δύο Ευρωπαίους πολίτες που κρατούνται στην Ινδία, μόνο αυτό που είπα μπορούμε να κάνουμε για να δοθεί προσοχή στην υπόθεση. Δεν είχα συγκεκριμένες προτάσεις από τους συναδέρφους, γι' αυτό εγώ προσπαθώ να φανταστώ από μόνη μου κάποιες λύσεις. Έχω στήριξη από ό,τι βλέπω από τους συναδέρφους, έτσι. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Και ελπίζω, αγαπητέ κύριε Στέφανο, το ταξίδι σας στις Βρυξέλλες να μην έχει γίνει για τίποτα. Να ξέρετε ότι εμείς δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, υπόθεσή σας και ευχόμαστε και εμείς θετική εξέλιξη για τους δύο αυτούς συμπολίτε μας, το μέλλον τους και τις οικογένειές τους να μεταφέρετε τις ευχές μας στις οικογένειες και τους φίλους, αν έχετε επαφή. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η αναφορά 0273 και 1177 από Ιταλούς πάλι Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στην, στον ε, αναφέροντα, τον κύριο Τζακόμο Ουτσιά, που είναι εδώ. Ε? Πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους για την ευκαιρία που μου δίνετε. Βρίσκομαι εδώ για λογαριασμό των πολιτών που έχουν τονίσει το τεράστιο πρόβλημα της ε, περιοχής του Λάτιου και της Ρώμης. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τα Μαρία Γκράτζια Βενούτη, η οποία ενεργοποίησε την αναφορά για την χωματερή της Μαλαγκρότα, που επρόκειτο να κλείσει από τον Οκτώβριο του 2013, αλλά ακόμα δεν έχει σφραγιστεί. Στην πράξη ε, γίνεται διήθηση στα υπόγεια ύδατα των αποβλήτων και λόγω εντόνων βροχοπτώσεων ε, μολύνει άμεσα και τα επιφανειακά ύδατα, το, το ποτάμια, τη θάλασσα, τον Τίβερη. Ε, τον Ιανουάριο του 2014 είδαμε να διαφεύγουν λίματα πέρα από την Μαλαγκρότα στις περιοχές που αφορούν τις γειτονικέ εγκαταστάσεις, δηλαδή είδαμε να υπάρχουν διαρροές και από τις εγκαταστάσεις της ΆΜΑ ε, για νοσοκομιακά λύματα, που είναι δηλαδή ειδική, ειδικός χώρος ταφής, ε, ρήπανση δηλαδή των ε, υπογείων υδάτων. Έχουμε στραφεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και στεραφήκαμε και στην, στο Πολυτεχνείο του Τωρίνου που έκανε έρευνα με μελετητές και τεχνικούς και προέβησε σχετική έκθεση. Παρ' όλα αυτά ο διαχειριστής δεν έχει ολοκληρώσει την προεκβολή της επιφανειακής σφράγισης της χωματερής ώστε να αποφευχθεί υπεραιτέρω περαιτέρω διήθηση ε, λιμάτων. Ο νόμος προβλέπει ότι οι πολίτες έχουν ήδη πληρώσει μέσω, από, μέσω των ε, τελών που έχουν καταβάλει για τριακονταετία και αυτό το ξεχνάνε οι τοπικές ε, αρχές. Ε, στην ουσία ο διαχειριστής έχει ζητήσει ένα είδος παράτασης λειτουργίας ε, της ε, χωματερής ε, μέσω ενός πόνους γιατί οι εγκαταστάσεις και οι δεντροφυτεύσεις που θα γίνονταν εκεί πριν το κλείσιμο θα κατέληγαν κατευθείαν να φύτευθούν πάνω στα λίματα. Ακόμα και τα τέλη που έχουν καταβάλει οι πολίτες είναι, είναι δυσανάλογα και αυτό το επιβεβαίωσε και το Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει εκδώσει απόφαση και την έχει γνωστοποιήσει στο Υπουργείο ε, Περιβάλλοντος. Εν τω μεταξύ ε, υπάρχει, αποφασι... φάνηκε ότι είναι λάθος το τέλος, είναι πολύ πιο ακριβό για τους πολίτες σε σχέση με αυτό που πραγματικά ε, θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί. Ε, Συνεχίζεται δηλαδή η ρήψη ευθυνών ανάμεσα στους ελεκτικούς οργανισμούς και τις τοπικές αρχές, οι οποίοι τελικά οι έλεγχοι γίνονται μόνο από ιδιώτες, όχι μόνο για τη Μαλαγκρότα, αλλά και για άλλες εγκαταστάσεις λιμάτων. Δεν γίνονται οι έλεγχοι, πάντα, ποτέ δεν έχουν λεφτά για ελέγχους, αλλά οι ιδιώτες μπορούν να διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις, να κάνουν τις business τους ωραία-ωραία και μετά να αφήνουν ε, ατελείωτα τα έργα. Υπάρχει και το πρόβλημα ε, των, ε, των εγγύσεων, των οικονομικών εγγύσεων, ώστε να μην πηγαίνουν κατευθείαν στην τσέπη τα χρήματα αυτού που είναι ο επιχειρηματίας. Αυτό επιτρέπει στο κοινό να μπορεί να υπάρχει εγγύηση σε περίπτωση που ο ιδιώτης ε, φύγει νωρίτερα, να ενεργοποιηθούν αυτά, αυτές οι εγκαταστάσεις όχι με δημόσια χρήματα, Γιατί εφόσον ο, ο επιχειρηματίας κερδίζει, θα πρέπει στο τέλος ο ίδιο να καλύψει και τι ζημιέ στο περιβάλλον. Όμως η αρχή αυτή του ορυπαίνων πληρώνει στην χώρα μας δεν γίνεται σεβαστή. Προσπαθήσαμε να έχουμε πρόσβαση για ορισμένες εγκαταστάσεις, αλλά και για τη Μαλαγκρότα ποτέ δεν μας επιτράφηκε, γιατί σύμφωνα με την περιφέρεια δεν υπάρχει πρόβλημα για το περιβάλλον. Οπότε εγώ διερωτώ με δεν έχουμε στοιχεία τα οποία είναι ευαίσθητα για τον ε, ιδιοκτήτη, γιατί αυτό επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα στο τέλος ζωής ε, του συγκατάστασης να πάρει κάποια επιδότηση. Πρόκειται για δράσεις οι οποίες ε, καλύπτονται απόλυτα από τη Σύμβαση Όρχους. Ζητάμε λοιπόν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρχει διαφάνεια Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι παρότι υπάρχουν απαγορεύσεις ε, και πρέπει να κλείσουν αυτές οι χωματερές, ζητείται από τους ιδιώτες με το νόμο 25 που σημαίνει απεμπλοκή, απεμπλοκή στην Ιταλία ε, να χρησιμοποιηθεί ένα μηχάνημα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Ιταλία. Ξεχνάμε όμως ότι γύρω από αυτή την ε, χωματερή υπάρχουν περιοχές σε Βέζο και ποτέ δεν έχει γίνει η παρέμβαση του δημόσιου τομέα εδώ και οι πολίτες ποτέ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν μπορέσει να συμμετάσχουν στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εγώ έχω δώσει τεκμηρίωση και σε σχέση με τα άλλα σημεία και τις άλλες ε, ε, αναφορές που αφορούν το Λάτιο, δηλαδή την χωματερή του Μόντε Ντελορτάτσιο που και εκεί εκκρεμεί απόφαση με αντίστοιχες επιπτώσεις και άλλες αναφορές ε, που αφορούν ένα σωρό άλλες, άλλους χώρους υγειονομικής ταφής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζουτζούσα. Το λόγο τώρα έχει η Επιτροπή για περαιτέρω διευκρινήσεις, αν αυτό είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο για να σας παρουσιάσω τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση, όσον αφορά τη διαχείριση λιμάτων στο Λάτιο. Μετά από την απόφαση του δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2014, η Κομισιόν παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση. Υπήρξε μια πρώτη επαφή με τις Ιταλικές Αρχές τον Μάρτιο του 2015 που αναφέρθηκε στην προηγούμενη μα ε, επικοινωνία με το Κοινοβούλιο και στη διάρκεια αυτή τη επαφή, οι Ιταλικέ αρχέ δεσμεύτηκαν να διαβιβάζουν περιοδικά στη Κομισιόν μια ενημέρωση όσον αφορά τι διαδικασίε αναθεώρησης των αδειοδοτήσεων των ε, χώρων υγειονομική ταφή του Λάτιου ώστε να ξέρουμε ότι, να επιβεβαιώνεται μάλλον ότι στις, ε, στους χώρους αυτούς μεταφέρονται λίμματα τα οποία έχουν υποστεί προτερή επεξεργασία Μάλιστα, οι Ιταλικές αρχές υποχρεώθηκαν και δεσμεύτηκαν ότι θα δίνουν ε, ε, πρακτικά για τις ενέργειες και τις δράσεις που γίνονται σε αυτές τις χωματερές. Αυτό επιβεβαιώθηκε τελευταία φορά το Φεβρουάριο του 2016. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν εξετάζει την ενημέρωση αυτή επί τη βάση της έκβασης αυτών των εκτιμήσεων, των αξιολογήσεων. Θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε ώστε να προχωρήσουμε στην κατάλληλη εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Ρέμο Ταβερνάρη από τη μόνιμη την προσωπία της Ιταλίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Μια σύντομη ενημέρωση. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Αναφορών για την πρόσκληση και άμεσα συνδέομαι με τα όσα είπε η συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ιταλικές αρχές έχουν ε, λάβει σε προηγούμενη συνάντηση το Μαρτίο 2015 διάφορες δεσμεύσεις και εμείς ως μόνιμη αντιπροσωπεία ζητάμε την αποστολή από πλευράς των αρμοδίων αρχών αυτών των ενημερώσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι να σας δώσω μια πρόβλεψη για την τελευταία ενημέρωση μετά από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, μια ενημέρωση που αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες, αν όχι μέρες. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν το Φεβρουάριο, ότι δηλαδή η διαδικασία για την έγκριση των χώρων υγειονομικής ταφής έχει στην ουσία ολοκληρωθεί η απόφαση της αναγνώρισης της περιφέρειας του Λατίου ήδη ανέφερε την ε, τύπης προσαρμογή όλων των εγκρίσεων που σχετίζονται με τους χώρους υγειονομικής ταφής, δηλαδή να διαγραφούν από τις προβλέψεις οι νομικές διατάξεις που επέτρεπαν την μεταφορά μη κατεργασμένων λιμάτων. Το Φεβρουάριο έμενε μόνο να προσαρμοστεί επισήμως η Αδειοδότηση για το ε, χώρο του Κόλεφα Φατσολάρα που εντωμεταξύ προσαρμόστηκε. Η επόμενη λοιπόν ενημέρωση θα σας δώσει τις, ε, τα στοιχεία της πράξης που επέτρεψε τη, επίσημα την προσαρμογή και της αυτής, ε, του τελευταίου αυτού χώρου Όσον αφορά το δεύτερο σημείο της απόφασης που είναι, θυμίζω, αυτή που δεσμεύει τις Ιταλικές αρχές στην εκτέλεση των όσων αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2014, δηλαδή τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαχείρισης των αστικών λιμάτων του της περιφέρειας του Λάτιου. Το σημείωμα που θα σταλεί τις επόμενες εβδομάδες θα επιβεβαιώσει την τάση που ήδη σημείωσαν οι εθνικές αρχές το Φεβρουάριο ε, του τρέχοντος, ότι δηλαδή οι δυνατότητες κατεργασίας των, των ε, αστικών λιμάτων για το 2016-2017 είναι πλέον επαρκής. Είχαμε το Φεβρουάριο 2016 στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Λάτιο είχε αναφερθεί η μηχανική βιολογική επεξεργασία του χώρου της Βιντόνια που αυτή τη στιγμή περιμένει την αδειοδότηση για να μπορέσει να λειτουργήσει και ελπίζουμε πως έτσι θα μπορέσουμε να ε, οδηγηθούμε και στη λειτουργία της ε, μονάδας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων της Γκουιντόνια. Θα δούμε έτσι ότι στο μέλλον οι μελλοντικές επιθεωρήσεις στους χώρους υγειονομικής ταφής θα δώσουν και προστιθέμενη αξία σε σχέση με την εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την απόφαση του Οκτωβρίου 2014. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχει έρθει η ώρα για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών. Ο κύριος Κοτσολίνο θα αρχίσει. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να ζητήσω μια πληροφορία όσον αφορά την, την, την, ε, τον νόμο σταθερότητας ε, του Σμπλοκ Ιτάλια. Όσον αφορά το ε, εργοστάσιο αερίου από λίμματα στην Μαλαγκρότα. Εδώ μιλάμε και τρέχουμε πίσω από τις πληροφορίες που μας στάνουν από τις διάφορες αρχές. Και μόλις σήμερα το πρωί ο τύπος λέει ότι η περιφέρεια η οποία έχει κληθεί από το κράτος να πει αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις ώστε να ξαναανάψει αυτή η μονάδα, έχει τελειώσει τις εργασίες της και είπε πως όχι δεν γινόταν να ξαναχρησιμοποιηθεί η λόγο ε, μονάδα. Άρα λοιπόν αναφέρον θα πρέπει να θεωρήσει ότι έγινε δεκτή η αναφορά του γιατί παρά τον νόμος Μπλοκα Ιτάλια, παρά τα όσα υπόθηκαν πριν, μετά από την, τον έλεγχο δεν δόθηκε η άδεια λειτουργία σε αυτήν την μονάδα. Εν μέρη λοιπόν οι τοπικές αρχές αντιμετώπισαν το πρόβλημα. Πώς να αρχίσω. Να αρχίσω με αυτό που είπε ότι το, δεν φταίει το μήνυμα, φταίει αυτός που το φέρνει. Μου φαίνεται πως όλα ε, πάνε καλά, ωστόσο πολλές φορές στην Επιτροπή Αναφορών έχουμε διαπιστώσει ότι η πραγματικότητα της επόμενης εβδομάδας είναι διαφορετική, ότι τα πράγματα δεν γίνονται όπως έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, ότι δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Εάν εφαρμόζονταν τότε όλα θα ήταν τέλεια, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, αν μπορούσαμε να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή, έτσι ώστε να λάβουμε πληροφορίες μετά από τον αναφερόμενο, ε, από τον αναφέροντα ότι έχει όντως γίνει αυτό που έχει προγραμματιστεί να γίνει, τότε θα ήταν ε, ίσως η καλύτερη λύση. Διότι πολλές φορές έχει συμβεί να χαιρόμαστε για την καλή μας δουλειά και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα από την άλλη πλευρά. Ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει και ο συνάδελφος σε αυτό. Εάν είστε 100% σίγουρος δηλαδή, τότε να κλείσουμε την αναφορά. μας. αν υπάρχει έστω και παραμικρός κίνδυνος, ας την αφήσουμε ανοιχτή. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε ΕΛΚ και σοσιαλδημοκράτε. Αλλά τώρα θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα. Για δύο λεπτά το πολύ. Για τις πληροφορίες στις οποίες αναφερθήκατε για τον αγγελιοφόρο, ε, για το μεσαντζέρο σήμερα το πρωί, αυτά είναι πληροφορίες, αλλά ε, η Περιφέρεια πήρε όλες αυτές τις πληροφορίες το τέλη του Μαρτίου. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτές τις πληροφορίες ε, από το Λάτιο, δηλαδή τόσο από την Περιφέρεια όσο και από την ε, πρωτεύουσα. Αυτά τα έχει λοιπόν στα χέρια της η περιφέρεια και όλο στοιχείως βγήκε και ένα άρθρο στον τύπο. Εμείς ε, δεν θέλουμε τέτοιου είδους αλλαγής γιατί η κέντρα εξουσία που μετακινούνται σε άλλα μέρη τη περιφέρειας του Λατίου τελικά δεν οδηγούν σε πραγματικέ αλλαγέ. Θέλουμε λοιπόν σιγά σιγά να συγκεντρώσουμε όλο το υλικό και να τεκμηριώσουμε με ουσιαστικό τρόπο αυτό που εμεί καθημερινά βλέπουμε. Δηλαδή ότι δεν είναι διαφανή η διοίκηση, η τοπική διοίκηση και οι πολίτε έχουν τεράστιε δυσκολίε να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με το περιβάλλον. Καθημερινά όποιο ξυπνά ε, έρχεται και λέει τα αντίθετο από ό,τι είπε την προηγουμένη. Πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να εμποδίσουμε τη λειτουργία, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό και καλό την Ευρώπη να παρακολουθεί από κοντά την τελεία για τη διαχείριση των λιμάτων. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα και ξεπερνάνε τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά και τις τοπικές αρχές και την πολιτική. Και αυτό το βλέπουμε εμείς καθημερινά. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει, να κρατήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά και να επαγρυπνεί έτσι ώστε ανα πάσα στιγμή να μπορεί να παρέμβει. Thank you very much. We now come Ευχαριστώ πολύ. Συμπερασματικά λοιπόν θα έχω να σας προτείνω το εξής. Καταρχάς αναγνωρίσουμε ότι έχετε το θάρρος αυτής της ανταλλαγής απόψεων. Αυτό που έχω να προτείνω στους συναδέλφους είναι να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή, να στείλουμε όμως μια επιστολή στις Ιταλικές Αρχές, να ζητήσουμε και από τον αναφέροντα να παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με την Επιτροπή η οποία διενεργεί συνεχείς αξιολογήσεις πρόοδου και όταν δούμε ότι σχεδόν έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, να μας στείλουν με τη σειρά τους μια επιστολή ότι όλα είναι υπό έλεγχο και όταν λάβουμε λοιπόν μια επιστολή και από τον αναφέροντα και από την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείσουμε την αναφορά, αλλά προς το παρόν να μείνει ανοιχτή. Πώς σα φαίνεται ο συμβιβασμό αυτό, Ωραία. Έτσι θα πράξουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι πίσω στην Ιταλία. Και είμαι σίγουρη ότι ο ήλιος σας φέρεται καλύτερα από ό,τι σε εμάς. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήρθατε και που παρακολουθείτε και θα παρακολουθείτε επάγρυπνα την κατάσταση. Περνάμε τώρα στο σημείο 25, αναφορά 18-18 και 18-19 από τον Μάθιου Τσάντερ για άδεια οδήγηση από τη Μάλτα που έπρεπε να αλλάξει σε Ιρλανδική. Ο κύριος Τσάντα δεν είναι παρόν, όμως μας έχει στείλει ένα μήνυμα μέσω βίντεο, το οποίο θα δούμε αυτή τη στιγμή. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών, θα ήθελα να ε, σας παρουσιάσω την αναφορά μου. Ε, αρχίζοντας με τη 18-18 2014 και 18-19 2014. Το σημείο δηλαδή 25 της ημερήσιας διάταξης που έχετε. πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που φέρνει τα κράτη-μέλη πιο κοντά στην Ευρώπη. Πολλές ε, περιπτώσεις έχουμε παρατηρήσει όπου στην Ευρώπη για χρόνια ολόκληρα σχεδιάζουμε νομοθετικά ε, πλαίσια τα οποία μετά παρακάμπτονται από ε, διάφορες εθνικές ρυθμίσεις και κοροϊδεύουν αυτό που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε, να χτίσουμε δηλαδή μια καλύτερη Ευρώπη. Η Οδηγία 2006-126 της 20 Δεκεμβρίου 2006 περιέχει το άρθρο 2 ε, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση αδειών οδήγησης. Η ουσία της οδηγίας αυτής δεν βασίζεται μόνο στο ότι όταν ταξιδεύεις ανάμεσα σε κράτη-μέλη μπορείς να χρησιμοποιήσεις την άδεια οδήγησή σου σε αυτά, αλλά πάει και παραπέρα διότι εάν ήταν έτσι τα πράγματα, σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έμπαιναν στον κόπο ε, να, ε, να δημιουργήσουν αυτόν τον ε, νόμο. Εάν ταξιδεύετε κι εσείς από εγώ, θα ξέρετε πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσεις την άδεια οδήγησή σου παντού στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία όμως δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό. Έχει φτιαχτεί έτσι ώστε οποιαδήποτε άδεια οδήγηση ενό κράτου μέλου να μέλους να ισχύει παντού. Οπουδήποτε δηλαδή στην επικράτεια της Ένωσης μπορεί κάποιος να οδηγήσει με άδεια οδήγηση άλλου κράτους μέλους. Και φυσικά είναι αυτονόητο ότι μπορείς να διατηρήσει την άδεια οδήγησή σου μέχρι αυτή να λήξει και μετά να την αντικαταστήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένεις. Και αυτό είχα σκοπό να κάνω όταν ε, μετακόμισα στην Ιρλανδία. Η άδεια οδήγησή μου της ε, Μάλτας έλεγε το 2020. Έτσι λοιπόν ε, δεν υπήρχε λόγος να αντικατασταθεί εφόσον δεν έλεγε ακόμα. Όμως στην Ιρλανδία υπάρχει διάκριση εις βάρος οδηγών που δεν κατέχουν Ιρλανδική άδεια οδήγηση. Και παρότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει ότι οποιαδήποτε άδεια οδήγηση κράτους μέλους πρέπει να αναγνωρίζεται, δεν ε, συνέβη στην περίπτωσή μου. Συμφωνώ πως χρειάζεται να γίνει μια εκτίμηση για το αν ο οδηγός πρέπει να λάβει την Ιρλανδική άδεια οδήγησης. Όμως ε, αυτό ε, πρέπει να γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και στα οποία δεν ανήκει η εθνικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Στις 22 Δεκεμβρίου 2015 έλαβα την απάντηση από την Επιτροπή ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν τα ασφάλιστρα ως εκείνα πιστεύουν αρκεί να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια καθώς και ε, να επιβάλλουν τις αντίστοιχες ε, ποινές. Όμως ε, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε σχέση με τον κώδικο δικής κυκλοφορίας και, τις, και τα πρόστιμα αλλά όταν γίνεται διαφοροποίηση των ετοιμών βασισμένη στην χώρα στην οποία της οποίας την κατέχει ο οδηγός, τότε αυτό κατα... καθιστά διάκριση. Στην Ιρλανδία λοιπόν, όταν πας να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου και δουν ότι, ανήκεις, ε, ότι η αδειοδήγησή σου έχει εκδοθεί σε άλλο κρατος τότε τα ασφαλίστρα είναι αυτομάτως ε, υψηλότερα και αν τους ρωτήσεις γιατί θα σου απαντήσουν ότι πρέπει να πληρώσεις περισσότερο ακριβώς επειδή δεν έχει Ιρλανδική άδεια οδήγησης. Μας κοροϊδεύουν. Και αυτό φαίνεται ε, στο ότι όταν αλλάξεις την άδεια σου και πάρεις την Ιρλανδική, τα ασφάλιστρα μειώνονται. Τι έγινε, έγινες καλύτερος οδηγός από τη στιγμή που πήρες την ε, Ιρλανδική άδεια οδήγησης. Δεν νομίζω. Μήπως είναι ένας έμεσος τρόπος φορολόγησης όλων των ε, πολιτών που φτάνουν στην Ιρλανδία και δεν θέλουν αυτόματα να αλλάξουν την άδεια οδήγησής τους και να πάρουν την Ιρλανδική θα έπρεπε να υπάρχει άμεση αναγνώριση των αδειών οδήγησης. Και να σας υπενθυμίσω ότι δεν ε, πρόκειται για θέμα αξιολόγηση του πόσο επικίνδυνο είναι ο οδηγό, διότι μπορώ να σα ε, απαριθμίσω πολλέ περιπτώσει όπου δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επιτρέπει ε, εθνικέ ρυθμίσει που παρακάμπτουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μην επιτρέπει να χρεώνονται υπήκοοι άλλου κράτους μέλους ε, μεγαλύτερα ποσά μόνο και μόνο επειδή είναι ξένοι στη χώρα αυτή. Είναι δίκαιο λοιπόν αυτό θα σας αφήσω να το αποφασίσετε εσείς. Η επόμενη αναφορά έχει σχέση με την ε, αλλαγή της αδειάς μου του διπλώματος οδήγησης σε Ιρλανδικό μέσα σε ένα ε, εύλογο χρονικό διάστημα. Να σας υπενθυμίσω ότι οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούσα να αλλάξω ε, το δίπλωμα οδήγησης ήταν αυτοί που προανέφερα. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κοιτάξει με προσοχή την αναφορά 18-18, διότι είμαι σίγουρος πως και εσείς ε, καταλαβαίνετε πόσο δυσάρεστο είναι να μην μπορείς να οδηγήσεις για μήνες περιμένοντας να ε, πάρεις το νέο σου δίπλωμα οδήγησης. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου έπρεπε να νοικιάσω αυτοκίνητα και αυτό κόστισε. Κόστισε αρκετά χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είχα καταβάλει εάν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Χρειάζεται να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για την ε, αλλαγή των ε, διπλωμάτων οδήγησης έτσι ώστε να αποφεύγονται τέτοιες, τέτοιες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ. Αναρωτιόμουν, λέει η Πρόεδρος, πόσο θα κρατούσε αυτό ακόμα. Αλλά εντάξει. Χάρη στον αναφέροντα, ο οποίο με ιδιαίτερα παιδαγωγικό τρόπο μας εξηγεί τι απόψεις του για την αναφορά αυτή, καταλάβαμε. Τώρα, η Επιτροπή, ο κύριος Λούκατ έχει το λόγο και ο κύριος Λίζη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στην, αναφορά 18-18-2014 και για την άλλη θα είναι ο συνάδελφος. Λοιπόν, όσον αφορά την ανταλλαγή αδειών οδήγησης, υπογραμμίζει ο αναφέρον ότι υπάρχει η αμοιβαία αναγνώριση βάσει οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις έγκυρες άδειες οδήγησης και ότι δεν χρειάζεται αυτές να ανταλλάσσονται εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν. Έτσι διασφαλίζεται το ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις και επίσης διασφαλίζεται και ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νομοθέτης αποφάσισε ότι εφόσον υπάρξει ανταλλαγή, οι χώρε μέλη είναι αρμόδιες για να αποφασίσουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται... γιατί δεν έχει την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει στις πρακτικές αυτές τη εθνικές ανταλλαγή. Όμω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες μέλη για να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται βέλτιστες πρακτικές και σε αυτές τις διαδικασίες ανταλλαγής διπλωμάτων οδήγησης και ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να υιοθετούν αποτελεσματικές πρακτικές. Αυτό γίνεται μέσω της Επιτροπής για τα διπλώματα οδήγησης που συστήνουν στις χώρες μέλη να ακολουθούν διαδικασίες οι οποίες δεν ε, εμποδίζουν τους οδηγούς να μπορούν να οδηγήσουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανταλλαγής. 27 Ιανουαρίου που μας ε, πέρασε είχαμε τα τελευταία δεδομένα και μπορούμε να επανέλθουμε αν θέλετε. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδήγησης ώστε ακριβώς η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των αρχών των χωρών μερών να μπορεί να γίνεται χωρίς ε, πρόβλημα και καθυστέρηση. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις χώρες μέλη λοιπόν για να διασφαλίσουμε ότι η οδηγία όσον αφορά τις άδειες οδήγησης θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά και ορθά στα πλαίσια πάντα της σημερινής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Θα προσθέσω λιγάκι όσον αφορά την ασφάλιση των οχημάτων. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Τσαντάουρ, δηλαδή ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να καθορίσουν την τιμολόγηση οι ίδιες. Δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση. Ούτε επιτρέπεται κάτι τέτοιο, ούτε καν σε επίπεδο χώρας μέλους. Τι κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αποφασίζουν ποιο είναι το προφίλ του οδηγού, του ασφαλισμένου και είναι ελεύθερες να επιλέξουν τα κριτήρια που θέλουν. Τώρα, κατά πόσο θεωρείται παράγοντας κινδύνου το από πού έχει εκδοθεί η άδεια οδήγηση. Η Μαλτέζικη άδεια οδήγηση δεν υποβάλλεται στο point system που ισχύει στην Ιρλανδία. Θεωρητικά δηλαδή εφόσον δεν υποβάλλεται στο σύστημα αυτό, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της οδήγησης, γιατί τότε έχεις λιγότερα κίνητρα, ας πούμε, να οδηγάς ασφαλώς. Εφόσον δεν υποβάλλεσαι σε αυτό το σύστημα. Άρα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα αντικειμενικό κριτήριο που ακολούθησε η ασφαλιστική εταιρεία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ωραία, πάει η Ιταλική Επιτροπή που είχα εδώ. Τώρα είναι πιο πολύ μαλτέζικη από ό,τι βλέπω βάσει συμμετοχή. Η Ρομπέρτα έχει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ Σεσίλια. Θα αρχίσω λέγοντας ότι κοίταξα την αναφορά αυτή και όλες τις αναφορές του κύριου Τσάνταρ και βάσει των όσων έχουμε από την γραπτή απάντηση της Επιτροπής και όσα μας είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Είδα ότι αναφέρεται το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδήγηση για να διευκολύνεται η ανταλλαγή διπλωμάτων οδήγηση μεταξύ των χωρών ε, μελών. Και η Μάλτα και η Ιρλανδία συμμετέχουν σε αυτό το ενωσιακό δίκτυο, είναι συνδεδεμένε. Χωρί όμω να κάνει αυτό καμία διαφορά. Γιατί 12 εβδομάδε έπρεπε να περιμένει ο κύριο Τσάντερ χωρί να μπορεί να οδηγήσει στο διάστημα αυτό. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι θα μπορούσε η ανταλλαγή αυτή να γίνει πιο εύκολα, πιο καλά. Το συμπέρασμα τώρα τη επιτροπή, ότι δεν υπάρχουν βάσεις για παρετέρω δράση είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη. Νομίζω ότι η ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κοιτάξουμε με περισσότερε λεπτομέρειε όπως και η βελτίωση του δικτύου αυτού αδειών οδήγηση. Γιατί στο κάτω-κάτω γι' αυτό υποβάλλουν αναφορέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πολίτε για να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Δεν μπορούμε εμεί να λέμε κάθε φορά ότι επειδή δεν υπάρχει η αρκετή αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε τίποτα, γιατί υπάρχει και εσωτερική αγορά στο κάτω-κάτω. Είναι θέματα και εσωτερική αγορά. Οπότε κύριε Πρόεδρε, ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και όταν επανέλθουμε το φθινόπωρο με θέματα εσωτερικής αγοράς εδώ στην Επιτροπή μας να ξανασυζητήσουμε και αυτό. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που σίγουρα δεν έχει μόνο ο κύριος Τσάντερ αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες ανά την Ήπειρό μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα εξετάσω και τις δύο αυτές αναφορές αυτό που λέει η Επιτροπή είναι λίγο αντιφατικά. Γιατί η ανταλλαγή αλλού γίνεται αποδεκτή χωρίς κανένα πρόβλημα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πιο ακριβά ασφάλιστρα και ότι δεν είναι επιλογή το αν θα ασφαλιστεί κανείς ή όχι, αυτό οδηγεί σε διάκριση. διότι επειδή αλλιώς θα χρεωθεί ακριβότερα ασφάλιστρα, οδηγείται ο ασφαλιζόμενος στην υποχρέωση να ανταλλάξει την άδεια οδήγησή του. Άρα δεν έχει την επιλογή, όπως λέτε. Καταλαβαίνω το εμπορικό επιχείρημα και εγώ έρχομαι από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνω ότι έχουν το προνόμιο ασφαλιστικές εταιρείες να αποφασίζουν για τα ασφαλιστρά τους, αλλά πιστεύω ότι χωρίς καμιά φιβολία ο πολίτης αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διάκριση που γίνεται εις βάρος του. Θα ήθελα να μείνει ανοιχτή λοιπόν η αναφορά αυτή και όχι μόνο για τον κύριο Τσάντερ, ο οποίος εδώ και μήνες έχει έρθει σε επαφή με το γραφείο μου και πολύ χαίρομαι που μπόρεσα να τον βοηθήσω να εμφανιστεί μπροστά μας, αλλά και προς όφελος άλλων πολιτών που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση και δεν έχουν κάνει αυτό που έκανε ο κύριος Τσάνταρ. Υπάρχει διάκριση σε βάρος των ε, πολιτών και αυτό ακριβώ είναι που θέλω να πω και να τονίσω. Γι' αυτό συστήνω να παραμείνει ανοιχτή παρακαλώ αυτή η αναφορά. Πρόεδρος, ωραία, τότε ολοκληρώνουμε ότι παραμένει ανοιχτή Α, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που πολύ σωστά είπε η συνάδελφος. Ναι, ναι, να την αφήσουμε ανοιχτή, όμως χρειαζόμαστε και κάποιες πληροφορίες. Γιατί δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία χρεώνει τόσο υψηλά ασφάλιστρα. Ναι, δηλαδή η απάντηση είναι ε, τους επιτρέπεται να το κάνουν αυτό, είναι για μένα πολύ απλή. Γιατί τους επιτρέπεται. πρέπει να μας εξηγήσουν το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν. Εντάξει, αν βασίζεται στον κίνδυνο που μπορεί να αποτελεί να οδηγό. εντάξει, αλλά έχω την ε, αίσθηση ότι δεν είναι μόνο αυτό. Διότι και ο αναφέρον ε, μας είπε ότι απευθύνθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία και τους είπε ε, δεν είναι δικό μας το θέμα κτλ. Πρέπει απλά να πληρώσετε. Δεν είναι αιτιολογία αυτή που χρησιμοποιήθηκε. Ναι, και εμένα μου φαίνεται πως είναι θέμα διάκρισης εδώ. Αλλά ίσως να υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να μην γνωρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Το έχω παρατηρήσει σε πολλά κράτη-μέλη. Όταν βρίσκομαι εκτός ε, Γερμανίας, ε, αντί να πάρω πόντους ε, για μια παράβαση, πληρώνω υψηλότερα πρόστιμα, ας πούμε, όπου δεν υπάρχει το ίδιο point system. Και εντάξει, μπορώ να καταλάβω το, την, ε, τις αρχές Ιρλανδίας, αλλά και πάλι δεν ε, έχω αρκετές πληροφορίες. Μάλιστα. Από ό,τι έχω καταλάβει, λοιπόν, πρόκειται για έναν υπήκο, Μαλτέζο υπήκο που μένει στην Ιρλανδία, και πληρώνει ασφάλιστρα 44% υψηλότερα από αυτά που πληρώνει ένας Ιλλανδός πολίτης για το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ε, αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή όπως είπαν και οι συνάδελφοι και να στείλουμε μια επιστολή στις Ιρλανδικές ε, αρχές στην ασφαλιστική, στην ασφαλιστική εταιρεία και να τους ζητήσουμε να μα δώσουν εξηγήσει ε, σχετικά με το γιατί έχουν χρεώσει περισσότερο τον άνθρωπο αυτό. Ε, μου φαίνεται πως ε, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε περίπτωση διάκρισης και εμπόδιο στην ελεύθερη μετακίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις λάβουμε απάντηση από τις Αρχές, θα τις προωθήσουμε στον αναφέροντα και θα κλείσουμε τότε την αναφορά. Διότι ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει λόγος ε, να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη αναφορά, αλλά δεν νομίζω πως ε, είναι τόσο απλό το θέμα. Ωραία. Ευχαριστώ. Το Σημείο 26 της σημερισής διάταξης. Εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος καμιά φορά ταξιδεύει και με αεροπλάνο. Γιατί πρόκειται για τον ίδιο αναφέροντα. Ο, ο αναφέρον είναι εδώ, πάλι με βίντεο, για να μας παρουσιάσει την αναφορά του. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Πέτη. Πρόκειται για την αναφορά 2032 του 2014 όσον αφορά την απαγόρευση αεροπορική εταιρεία επιβίβαση κατοικιδίων ζώων στην καμπίνα επιβατών. Είναι μια απόφαση μονομερής της εταιρεία. Όμως πλήττει μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω την περίπτωσή μου για να καταλάβετε σαφώς το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω. Έχω ένα μικρό κατοικίδιο ζώο, αμυνιατούρα θα έλεγα, πολύ μικρό, το οποίο έχει το μέγεθος ε, που θα μπορούσε κάλλιστα να ταξιδέψει στην καμπίνα επιβατών. Όμως αυτό μπορεί να συμβαίνει παντού, εκτός από την περίπτωση της Ιρλανδίας. Εμείς μετακομίσαμε στην Ιρλανδία πριν από τρία χρόνια και επειδή χρειαζόμασταν αυτοκίνητο, πήγαμε με αυτοκίνητο από τη Μάλτα στην Ιρλανδία με το σκυλάκι μας στο αυτοκίνητο. Και επειδή αρέσει πολύ στη σκελίτσα μας να ταξιδεύει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και φτάσαμε μέχρι την Ιρλανδία χωρί κανένα πρόβλημα. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα με το αεροπλάνο. Γιατί αν προσπαθήσετε να φύγετε από την Ιρλανδία με το σκυλάκι σα στην καμπίνα επιβατών, κανένα πρόβλημα. Για να επιστρέψετε όμω, δεν μπορείτε. Για μένα αυτό μου φαίνεται φοβερό. Καλέσαμε τη Λουφτχάνσα και μα είπαν ότι η Ιρλανδία και θεωρείται ως μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε έπρεπε να έρθω σε επαφή με το Υπουργείο Γεωργίας ε, για να πάρω την απάντηση στην κυρία Wells στις 13 Αυγούστου 2014 που είπε ότι είναι υποχρεωτικό να κατα... οι καταγραφόμενες αεροπορικές εταιρείες εκ των προτέρων να έχουν ενημερώσει για τα ζώα τα οποία θα καταλήξουν στην επικράτεια και ότι τελικά αποφασίζει κατά περίπτωση η ίδια αεροπορική εταιρεία. Αυτό όμως πρέπει να το συμπληρώσουμε το εξή. Η γυναίκα μου και εγώ είχαμε το πρώτο μας παιδί τον Ιανουάριο και αποφασίσαμε να περάσουμε δύο μήνες στην Μάλτα. Οπότε θελήσαμε φυσικά να πάρουμε και τη σκλίτσα μας μαζί. Στις 23 Μαρτίου ταξίδεψα με την Λουφτχάνσα μέσω Φραγκφούρτης και μετά με την Air Malta έφτασα στη Μάλτα με το σκυλάκι πάρα πολύ ωραία και στις δύο πτήσεις μαζί μου στην καμπίνα. Και συναντήθηκα με έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας της Μάλτας στο αεροδρόμιο και μου επέτρεψε αφού προηγουμένως ε, ήλεγξε ότι έχει εμβολιαστεί ο σκύλος λοιπά. Να εμπώ με το σκυλί μου στη Μάλτα. Τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε τον Ιούλιο στο Δουβλίνο. Δεν θα είναι εύκολο ταξίδι γιατί δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την αντίστροφη πορεία γιατί η Λουφτχάνσα δεν επιτρέπει να πάρουμε το σκελί μαζί μας στην καμπίνα επιβατών. Οπότε τι θα κάνω, θα πρέπει να πάω με την Air Malta και το σκυλί μέχρι το Παρίσι, να νοικιάσω αυτοκίνητο από εκεί, να ταξιδέψω μέχρι την άκρη της Γαλλίας στο Ροσκόφ, έξι ώρες δηλαδή, και μετά να πάρω ένα φεριμπότ για το Κόρκ ή το Ρόσλερ που θα μας κρατήσει περίπου 14 ώρες ε, στο ταξίδι. Και μετά να βρω έναν τρόπο να φτάσω στο Δουβλίνο. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να φτάσω στον προορισμό μου με τη σκυλίτσα μου. Είναι ένα σίτσου και έχει πλακουτσωτή φάτσα, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές ε, συνθήκες και να, δυσκολεύει, και να δυσκολεύεται η αναπνοή σε κάποιες περιπτώσεις. Κάτι το οποίο γνωρίζουν οι αεροπορικές εταιρείε που εκδίδουν και σχετικές οδηγίες. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι στην καμπίνα μαζί μου. Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, αν πραγματικά πιστεύει στην ευημερία των ζώων, θα έπρεπε να διασαφηνίσει το ζήτημα αυτό. Εδώ παίρνει αποφάσεις για άλλα θέματα, όπως είναι η κλωνοποίηση, που είναι στο κάτω-κάτω και λιγότερο ξεκάθαρο. Και είναι θέμα ελευθερίας ε, κυκλοφορίας της οικογένειας μαζί με το σκυλί τη. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Λουφτχάντσα λέει ότι μεταφέρει κατοικίδια το Υπουργείο Γεωργίας επίσης ε, έχει αποφανθεί όσον αφορά την ε, μεταφορά και την άφηξη ζών στην Ιρλανδία. Εδώ λέτε επίση καμιά φορά ότι είναι εμπορική πρακτική και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όμω για το roaming έχετε κάνει, έχετε πείσει τι επιχειρήσει να μειώσουν το κόστο. Έτσι θα έπρεπε να γίνει και με τι αεροπορικέ εταιρείε και να επιτρέπετε το ταξίδι των κατοικιδίων στην καμπίνα επιβατών σε όλου του προορισμού που βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σα και το σκληρό σα έργο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Μου φαίνεται αστείο, λέει η Πρόεδρος. Αλλά δώστε μας μια εξήγηση παρακαλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε δύο στάδια εξετάζουμε το θέμα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ομοθεσία αεροπορικών μεταφορών. Και μετά θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο για το θέμα υγείας των ζώων, που επίσης αναφέρεται εδώ. Λοιπόν, όπως λέμε και στην απάντηση που στείλαμε στον κύριο Σιάνταρ, δεν υπάρχει νομοθεσία σήμερα σε κοινοτικό επίπεδο που να ρυθμίζει την μεταφορά κατοικιδίων ζώων στην καμπίνα επιβατών ή μαζί με τις αποσκευές. Υπάρχει κάποια νομοθεσία, δύο μάλιστα, που θα μπορούσε να καλύπτει το θέμα. Το ένα είναι η ευθύνη σε περίπτωση κάποιας ζημιάς, βάσει της σύμβασης του Μόντρεαλ που έχει ενσωματωθεί στο κοινοτικό δίκαιο από το 1997 και υπάρχει και νομοθεσία η οποία καλύπτει το δικαίωμα των ατόπων μόνο με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα και που πρέπει να συνοδεύονται από ένα ζώο που τους βοηθάει στη μετακίνησή τους. Τότε βέβαια οι φυτογενομικοί κανόνες της κάθε χώρας πρέπει να τηρούνται πλήρως. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως λοιπόν έχουμε πει στον αναφέροντα, πιστεύουμε ότι σε επίπεδο ροπορικών μεταφορών Αν μπαίναμε στο νομοθετικό ζήτημα θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολλούς παράγοντες, το βάρος, το μέγεθος, ε, ένα σωρό παράγοντες σχετικά με το ζώο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει αρμοδιότητα ούτε και νομοθετικό σχέδιο, ούτε σκοπεύουμε να καλύψουμε αυτό το τομέα που κατά τη γνώμη μας είναι εμπορική απόφαση των αεροπορικών εταιριών που μπορούν να αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν ή όχι την πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα που συνοδεύουν έναν επιβάτη στην καμπίνα των επιβατών. Ο επιβάτης δεν έχει παρά να διαλέξει την ε, εταιρεία εκείνη η οποία έχει πιο ευνοϊκούς κανόνες όσον αφορά τη μεταφορά αυτή. Πρόεδρος. Ωραία. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο από τους βουλευτές. Α, ναι. Ακριβώς, συγγνώμη. Η κυρία Λάιν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλημέρα. Όσον αφορά την υγεία των ζώων, ο αναφέρον λέει ότι δεν ανταποκρίνεται στον κανονισμό του 2005 η αεροπορική εταιρεία. Το, η ρύθμιση αυτή μιλάει για τη μεταφορά ζώων εφόσον αυτή συνδέεται με μια οικονομική δραστηριότητα. Ενώ εδώ δεν πρόκειται για τέτοιου είδους μετακίνηση. Βέβαια θέλω να προσθέσω και το εξή. Η μετακίνηση των κατοικιδίων μεταξύ χωρών μελών ρυθμίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν πρόκειται για μη εμπορική μετακίνηση ή εμπορική, για το σκέλος που αφορά την υγεία τους. Οι χώρες μέλη, λοιπόν, πρέπει να διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται τα ζώα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Ιρλανδία, λοιπόν, από αυτού αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα του κανονισμού 80 του 84 που της επιτρέπει τον έλεγχο των κατοικιδίων αυτόν να τον αναθέσει σε οργανισμούς που εγκρίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον μεταφορέα, στην αεροπορική εταιρεία δηλαδή, γιατί η Ιρλανδία πιστεύει ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι περισσότερο σε θέση να ελέγξουν τα κατοικίδια όταν αυτά μπαίνουν στη χώρα. Οι μεταφορείς λοιπόν είναι επιτετραμένοι από τη χώρα από την Ιρλανδία να κάνουν τον έλεγχο αυτό. Και για τους μεταφορείς μία προϋπόθεση είναι ότι είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν την άφηξη των ζών 24 ώρες νωρίτερα με email στο, στην ιστοσελίδα της Ιρλανδίας που είναι μια συγκεκριμένη εκεί πρέπει να γίνει η κοινοποίηση στα πλαίσια αυτά λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο μεταφορές μπορεί να απαιτήσει το κατοικίδιο να μεταφερθεί όχι στην καμπίνα των επιβατών, αλλά μαζί με τις αποσκευές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα οι συνάδελφοι έχουν τον λόγο. No Ουδής. Καλώς. Περίεργο. Συνήθως Μιλάτε πολύ. Τι έγινε. Έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, διαβεβαιώνουμε τον ε, αναφέροντα ότι μπορεί να γελάσαμε γιατί ήταν η πιο ευχάριστη αναφορά αν θέλετε το να ταξιδεύεις με το ζωάκι σου έχει μια ανθρώπινη διάσταση οπότε γι' αυτό υπήρξε κάποια ευθυμία γιατί δίνει μια πραγματικά ανθρώπινη διάσταση <laughs> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε λοιπόν ότι δεν υπάρχει νομική βάση προκειμένου να παρέμβει, ότι είναι εμπορική φύσεως απόφαση αυτή από τους μεταφορείς. Και η ρύθμιση του 2004 για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά τους δεν εφαρμόζεται εδώ. Γιατί δεν πρόκειται για οικονομικό κέρδος με τη μεταφορά αυτή. Οπότε η αεροπορική εταιρεία είναι αρμόδια η Lufthansa στη συγκεκριμένη περίπτωση και είναι ελεύθεροι να ε, θέσουν τους δικούς τους κανόνες. Και λοιπά και λοιπά. Αυτό που έχω να προτείνω λοιπόν είναι να κλείσουμε την ε, αναφορά. Δεν υπάρχει νομική βάση για να υποχρεώσουμε τις αεροπορικές εταιρείες να εναρμονίσουν ε, τις ε, διατάξεις τους, τις πολιτικές τους μάλλον περί κατοικίδιων. Ε, είναι πιστική η επιχειρηματολογία, ωστόσο, και μπορούμε άμεσα να έρθουμε σε επαφή με τη Lufthansa και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε να κινηθούν προς τη δική μας κατεύθυνση. Εντάξει, ωραία. Και τώρα πάμε στην αναφορά. Ε, που αφορά την παραγωγή κίτρου εσπεριδοειδών βασικά. Πρόκειται για την υπαριθμόν 067. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ, αλλά παρακολουθεί την ε, συνεδρίασή μας που δίδεται ε, στο διαδίκτυο και τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Χεζούς Μεντέρο Μαρτίνες. Πρόσωπο της Επιτροπής. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χεσούς Μενέρο Εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας στο τμήμα των άμεσων πληρωμών και σε σχέση με αυτή την αναφορά θέλω να αναφερθώ στις παρατηρήσεις που παρουσίασε η Κομισιόν και που ακολουθούν την ίδια γραμμή με τη γνωμοδότηση που εξέδωσε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να θυμίσω λοιπόν ότι μετά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τελευταία στην κοινή γεωργική πολιτική δεν υπάρχουν πληρωμές οι οποίες να δεσμεύονται για συγκεκριμένους τομείς. Η μοναδική δυνατότητα επιδότησης ε, συγκεκριμένων τομέων αυτή τη στιγμή περιλαμβάνεται στο άρθρο 52 του κανονισμού 1307 ε, είναι το σύστημα των εθελοντικών δεσμευμένων ε, ε, πληρωμών και περιορίζεται σε κάποιους τομείς μεταξύ των οποίων είναι και τα φρούτα και λαχανικά Άρα και ο τομέας των εσπεριδοειδών. Σε για αυτούς τους λοιπόν υπάρχει δυνατότητα ε, τα κράτη-μέλη να προβούν σε συνδεδεμένες ενισχύσεις εντός του όριου που ισχύει για τέτοιου πληρωμές και για κάθε κράτος μέλος από τη στιγμή που πληρούνται κάποιοι όροι και προϋποθέσεις και το, περιλαμβάνονται αυτά στις δύο γνωμοδοτήσεις που σας δώσαμε. Πρέπει αυτοί οι τομείς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες εντός συγκεκριμένων ορίων και άρα λοιπόν κάθε κράτος μέλος είναι αυτό το οποίο αποφασίζει σε ποιους τομείς είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν αυτού του είδους οι πληρωμές στην Ισπανία όταν ξεκίνησε αυτό το σύστημα δεν συμπεριλήφθηκε ο τομέας των ε, φρούτων και πορκεπευτικών στο σύστημα ε, αλλά ούτε και τομέα των εσπεριδοειδών στους επιδοτούμενους τομείς. Θέλω να θυμίσω επίσης ε, ότι αυτά τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει η Ισπανία σε σχέση με τις ε, ε, δεσμευμένες ε, πληρωμές φέτος θα αναθεωρηθούν, θα επανεξεταστούν, θα ολοκληρωθούν δηλαδή πληρωμές για τους συγκεκριμένους τομείς και θα τροποποιηθούν ή θα συνεχιστούν και ή θα δοθούν σε νέους τομείς. Το Ισπανικό κράτος αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτές τις, αυτά τα μέτρα σε νέους τομείς, εάν το επιθυμεί. Άρα λοιπόν θεωρητικώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα αν είναι αλήθεια πως αυτοί οι τομείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διευθυντικά προβλήματα και χρειάζονται συγκεκριμένη ενίσχυση. Αυτή είναι η μοναδική δυνατότητα που υπάρχει, διότι δεν εξαρτάται από την Κομισιόν πλέον, αλλά από το το κράτος μέλος που επιλέγει τον τομέα αυτόν ως τομέα που αντιμετωπίζει δυσκολία και πρέπει να στηριχθεί. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ απλά θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους πριν σας δώσω το λόγο Πίτερ ότι πρόκειται για μια αναφορά την οποία εξετάσαμε στη διάρκεια της ε, άσκησης που είχαμε για την ε, εξέταση και λοιπόν στην Κομισιόν και ζητήσαμε περαιτέρω γνώμη και κατά τη γνώμη μου μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά αφού λάβαμε τις απαντήσεις που ζητήσαμε. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Θέλεις το λόγο Πίτερ πάλι. Όχι, πολύ καλά συνοψίσατε την αναφορά. Ίσως θα ήθελα να πω στον ε, αναφέροντα ότι η αναφορά του θα έπρεπε να απευθυνθεί όχι εδώ αλλά στην Ισπανία, στις Ισπανικές αρχές, ε, διότι μου φαίνεται πως εκεί βρίσκεται ο αρμόδιος. Είναι ένα θέμα αρκετά ε, αμφιλεγόμενο οι άμεσες ενισχύσεις, όμως πιστεύω πως ε, μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά και να κινηθούμε ήσυχοι, διότι ο αναφέρον θα πρέπει να απευθυνθεί στην ε, Ισπανική κυβέρνηση, στις Ισπανικές αρχές. Όπως ακούσαμε, αυτή η απόφαση μπορεί να λαμβάνεται εκ νέου μια, κάθε χρόνο, οπότε είναι στο χέρι των Ισπανικών αρχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει περάσει η ώρα, ασχοληθήκαμε με όλες τις αναφορές στην ημερήσια διάταξη και αυτή η μαραθώνια συνεδρίαση που άρχισε χθε της Επιτροπής Αναφορών έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε. Ε, ευχαριστώ πολύ στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Γραμματεία, σε εσάς, τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τους διερμηνείς. Συνήθως σας ζητώ 10 λεπτά παραπάνω, σήμερα όμως όχι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.